Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Νομίζω πως το μας, το χθεσινό μας κοκτέιλ, το ποτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήρθαν όλοι οι πιο σημαντικοί υπουργοί γεωργίας, ακόμα και αν ε, το ποτό που προσφέραμε ήταν ε, κάτι πολύ φτωχό. Σύμφωνα με τον προπολογισμό της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε κάτι πιο πλούσιο. Ε, ωστόσο, ακούσαμε εκτιμήσεις όλων των ε, Υπουργών. Να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Λούλινγκ για την σημαντική συνεδρίαση που έκανε για τον Ίνο. Υπογράμμισε αυτό το ρόλο της Κομισιό μας, της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου γενικότερα. Αν έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Σημείο 7. της ημερήσιας διάταξης. Εφαρμογή τη διμερού ρήτρα διασφάλιση και του μηχανισμού σταθεροποίηση για τι μπανάνε στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κολομβία και Περού. Ε, συγγνώμη, Κεντρική Αμερική, με συγχωρείτε. Ο κύριο Μαντρόβερ. Ε, να του δώσω γρήγορα το λόγο για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πραγματικά όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Ο Πρόεδρος ε, χτες αναφέρθηκε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, εγώ δεν μπόρεσα να δεχτώ όλες τις τροπολογίες. Πολλές από αυτές είναι λογικές, αλλά τροποποιούν την εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό μιλάω για τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου. Έτσι κι αλλιώς όταν ζητείτε γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ συχνά αυτό γίνεται αργά. Και γι' αυτό και δεν μπορούσα να δεχτώ τέτοιες τροπολογίες που είναι σε αντίθεση με τις συμφωνίες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ Καμπρίελ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και είστε όλοι έτοιμοι με τον κατάλογο ψηφοφορίας, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, να δούμε ότι ο αντιπρόεδρος Μποβέ δεν έχει την κάρτα του. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 21, πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα του άρθρου 21. Άρχεται η ψηφοφορία, είμαστε όλοι υπέρ. Ωραία, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για τροπολογία 7 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ωραία. 22 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22. Απορρίπτεται. 23 τώρα. Το εισηγητή. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 24. Θα λέω ότι απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την 25. 25 απορρίπτεται. Εννέα τώρα του εισηγητή ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 10 του εισηγητή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 του εισηγητή υπέρ, ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε για την ε, τροπολογία 12, τέλος της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 του εισηγητή, ψηφίζουμε, τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 26 τώρα. Είμαστε όλοι κατά, οπότε απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε κάποια εκτιμώντας. Μπορούμε να ψηφίσουμε unblock από το 14 έως και το 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Ποια να βγάλουμε, όλες, μία-μία. Allora che facciamo? Da 14 a 18. Siete d'accordo nel votare in blocco? Συμφωνείτε να ψηφίσουμε un blocco από τη 14 έως και τη 18? Συμφωνεί. No? Ok, allora andiamo avanti. Uh, numero 14. Όχι. Ωραία. Τότε προχωράμε. 14. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2 του εισηγητή. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρία του εισηγητή. Εγκρίνεται. πέντε Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεκαέξι. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 4. Το εισηγητή. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ταραμπέλα. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 19. 19 ποιος απέχει, ο Ταραμπέλα. 19, Μάτω. Εγκρίνεται. 5. Μα 5 τίποτα. 20 άλβες. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τοποποιήθηκε. Και εγκρίνεται συγχαρητήρια στον συνάδελφο Γκαμπριέλ. Να περάσουμε άμεσα στην επόμενη ψηφοφορία. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 8. Πάλι είναι ο εισηγητής ο Γκαμπριέλ Ματοδρόβερ. Είναι η εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης και το μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες ε, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας και Περού. Έτοιμοι όλοι. Ξεκινάμε την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Τροπολογία 6 εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 21 στο Γιανόφ. Άρχεται η, τροπο... η ψηφοφορία για την 21. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 22. Πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα της 22, όπου Είμαστε υπέρ. Τώρα ψηφίζουμε την 7 του εισηγητή. Εγκρίνεται. 23. Προσοχή 23. 23 ψηφίζουμε Νομίζω πως υπάρχει πλειοψηφία κατά. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην... Ψηφίζουμε για την 24. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 28. Την 25 ψηφίζουμε και τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην 26. Ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. Respinto. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 9. Aperta la votazione 9 του εισηγητή. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 10 του εισηγητή. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορία. εγκρίνεται. 11 του εισηγητή. Έγκρινεται. 12 του εισηγητή. Εγκρίνεται. 13 του εισηγητή. εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την 27. Ψηφίζουμε για την 27. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα σε τηλογικές σκέψεις. Chiedo Ψηφίζουμε για την εκτιολογική σκέψη 14. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1 λοιπόν υπέρ. Ε, ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε εγκρίνεται. 2 τώρα. Ψηφίζουμε για την δύο. 2. Αιτιολογική σκέψη του εισηγητή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 15. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Υπέρ. Εγκρίνεται. 16. Ψηφίσουμε για τη 16. Μεγάλη πλειοψηφία υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του εισηγητή. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 εγκρίνεται 18 ταραμπέλα μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του Μάρκ Ταραμπέλα πάντα υπάρχει ένας που απέχει πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός όχι ο Μποβέ δεν δεν έχει καν την κάρτα εγώ υπερψήφισα δεν είμαι εγώ Λοιπόν, 19 τώρα. 19 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 5 του εισηγητή. Όχι, 5 δεν την ψηφίζουμε. 20. Λουίς Αλβέσ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. εγκρίνεται σε χαρακτήρια, Γκαμπριέλ. Μπράβο. Πάμε στο σημείο 9. Προϋπολογισμός 2013. Εντολή για τον τριμερή διάλογο. Έχουμε την κυρία Έστερ Δελάνζ και είναι παρόν και ο κύριος Τζοβάν Λαβία που είναι γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2013. Η Επιτροπή μας έχει εδώ παρόντα τον Γενικό Εισηγητή επί του προϋπολογισμού. Όπως είχε γίνει και πέρυσι, η για το 2012 και ο κύριος Λαβία έχει σκοπό να κρατήσει στενή επαφή με τις ε, μεμονωμένες επιτροπές από την αρχική φάση της σύνταξης του προπολογισμού. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις πιθανές ε, προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2013 πριν ακόμα από την παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού από πλευράς ε, της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ένα σχέδιο προπολογισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα υποβληθεί στις 25 Απριλίου. Ε, να σας θυμίσω ότι αυτή η έκθεση ορίζει την εντολή της Επιτροπής Προϋπολογισμού για τον τριμερή διάλογο. Θα υποβληθεί στην Επιτροπή στις 10 Μαΐου και η υποβολή των τροπολογιών προβλέπεται για τις 31 Μαΐου και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού στις 20 Ιουνίου. Άρα θα περάσει από την Ολομέλεια κανονικά τον επόμενο Ιούλιο. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Βλέπω εδώ ο κύριο Λόγκο, διευθυντής και ε, το επιτελείο του είναι παρόντες. Να δώσω αμέσω ε, το λόγο στον κύριο Λαβία. Grazie, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως Ξέρετε, η διαδικασία η δημοσιονομική είναι μια μακρά διαδικασία. κρατά όλη τη διάρκεια του έτους και ε, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών που ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία στην Σύνοδο της Ολομέλειας του Στρασβούργου την περασμένη εβδομάδα. Έχω επισκεφθεί την Επιτροπή σας για πολλούς και διάφορους λόγους, εκτός από το ότι είμαι μέλος της Επιτροπής. Στόχος μου είναι να έχω μια στενή συνεργασία με όλους τους ε, ειδικούς ε, ε, εισηγητές, έτσι ώστε να κάνουμε μαζί την πορεία για την, μέχρι την έγκριση του προπολογισμού και να εντοπίσουμε ξεχωριστά ποιες είναι οι προτεραιότητες μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κάθε επιτροπής. Θα ήθελα να σας θυμίσω πως φέτος είναι η τελευταία χρονιά των δημοσιονομικών προπτικών για την περίοδο 2007-2013 και επειδή πρόκειται για την τελευταία χρονιά είναι ταυτόχρονα το έτος όπου τείνουν να συγκεντρώνονται όπως ε, ήθιστε στο τέλος κάθε προγραμματικής περίοδου οι ανάγκες πληρωμών. Για τον γεωργικό προπολογισμό η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική γιατί συμπίπτουν συνήθως οι υποχρεώσει με τις πληρωμές και δεν ε, προβλέπονται ίδιες δυσκολίες που υπάρχουν σε άλλα πλαίσια και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω ότι αυτός ο υπερπολογισμός ακολουθεί την συνδιαλλαγή για την ολοκλήρωση του προπολογισμού, το κλείσιμο μάλλον του προπολογισμού του 2012 που ήταν μια ιδιαίτερη χρήση για τον προϋπολογισμό. Το Συμβούλιο ε, αντιστάθηκε σε μια αύξηση των κονδυλίων για τις πληρωμές και λόγω της κρίσης ε, που φυσικά χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή και ε, περικόπτει εντόνως τους εθνικούς προπολογισμού και οδήγησε στο τέλος του περασμένου έτους σε μια πολύ, ε, ένα πολύ έντονο αίτημα για εκταμιεύσεις πληρωμών. Να φανταστείτε ότι μόνο το Δεκέμβριο του 2011 ε, τα αιτήματα αυτά έφτασαν στα 16 δις ευρώ, ενώ υπήρχαν στο Ταμείο διαθέσιμα μόνο 5 δις στο Ταμείο. Αυτό καθόρισε εν γέννη μια έντονη ανάγκη για πληρωμές που μεταφέρθηκαν στο προπολογισμό του 2012 και που προφανώς θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαδικασία προετοιμασίας για τον προπολογισμό του 2013. Στις κατευθυντήριες γραμμές που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια εστιάσαμε την προσοχή μας σε δύο προτεραιότητες. Από τη μια πλευρά ανάπτυξη και ανάκαμψη και δεύτερη ο σπηλώνας η απασχόληση με την εστίαση στο ε, επίλυση ενός προβλήματος που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα ε, και σε πολλά κράτη-μέλη συγκεκριμένα στην ε, ανεργία των νέων όπου σε κάποιες χώρες έχει ξεπεράσει ένα εξαιρετικά ψηλό επίπεδο που είναι το 40%. Ε, επίσης ε, θελήσαμε να τονίσουμε πως το 85% της νέας απασχόλησης των νέων θέσεων έχει δημιουργηθεί μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γι' αυτό και θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον προπολογισμό στις μικρομεσαίες γιατί ακριβώς θεωρούμε πως οι μικρομεσαίες είναι ένα στρατηγικό στοιχείο για την οικονομική ανάκαμψη και για την απορρόφηση του υψηλού επίπεδου μη απασχόλησης ανεργίας που χαρακτηρίζει πολλές χώρες. Όπως έλεγε και προηγουμένως ο Πρόεδρος, τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση για την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Και θα ήθελα να εδώ οι μεμονωμένες επιτροπές να κάνουν μια συζήτηση για το ποιες θεωρούν ότι θα είναι οι προτεραιότητες τους και όσα θα θέλουν να τις τονίσουν αυτές, αλλά και ποια είναι τα προγράμματα ή γραμμές του προπολογισμού που θεωρούν λιγότερο σημαντικές. Γιατί σε μια περίοδο κρίσης όπου θα πρέπει να εγκρίνουμε σίγουρα έναν λιτό προϋπολογισμό. Ναι, θα πρέπει να εντοπίσουμε τις προτεραιότητές μας, αλλά να δούμε και αν υπάρχουν και γραμμές προϋπολογισμού που δεν δαπανώνται, που οι προγράμματα τα οποία δεν είναι προτεραιότητες ή αρνητικές προτεραιότητες όπως τις αποκαλέσαμε. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι ακόμα πριν να κλείσω. Για μια άλλη ε, συνήθη προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσει. Για τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει θα έχουμε ένα πιο ειδικό χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε από την Εκτελεστική Επιτροπή μια, μια αρχική εκτίμηση για τη δυνατότητα ε, εκτέλεσης των συγκεκριμένων δράσεων. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε από τις μεμονωμένες επιτροπές, τις ειδικευμένες επιτροπές, να αναγνώσουν από κοινού μαζί μας ε, τις προτάσεις αυτών των, προτα... των πιλωτικών και προπαρασκευαστικών δράσεων που θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι τα τέλη Μαΐου από όλε τι επιτροπέ ώστε να διαβεβαστούν έπειτα στην Επιτροπή Προπολογισμού που στις 4 Ιουνίου θα στείλει το πακέτο αυτό των προτάσεων πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων στην Κομισιόν, ώστε εκείνη να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατόν να εκτελεστούν και θα μας στείλει πίσω την αναδιατύπωση. Να μας πει δηλαδή αν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, αν καλύπτονται ήδη από τις γραμμές του προπολογισμού και αν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν ή όχι. Μετά από το καλοκαίρι θα μπορέσουμε να τα τροποποιήσουμε, αν χρειάζεται τροποποίηση, ανάλογα με τις υποδείξεις που θα μας κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή και να φτάσουμε έτσι σε ένα τελικό πακέτο που θα είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων ε, που θα γίνουν ε, με τη συνδιαλλαγή μέχρι τον Νοέμβριο για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό στα τέλη Δεκεμβρίου ως ήθιστε. Ευχαριστώ πολύ ωραία. Ευχαριστώ ε, Τζοβάνι. Πρώτα η κυρία Ντελάνγκε. Ντελάνγκε πρώτα, φυσικά. Ναι. Όχι, ξέρω ποια είναι η θέση μου, μιλήσει πρώτα ο Γενικός αλλά μετά ίσως θα πρέπει και ο συγκητής της ε, Γεωργικής Επιτροπής να λάβει το λόγο. Αν και με βέβαια ότι και με τους κοιόδες συγκητές έχουμε, θα έχουμε καλή συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστώ λοιπόν τον Τζοβάνι Λαβία που είναι εδώ και Καλό είναι που έχουμε φέτος ένα γενικό εισηγητή που γνωρίζει καλά τα γεωργικά θέματα. Ξέρω ότι δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Είμαι ευγνώμων λοιπόν για την ε, παρουσία του εδώ και ξέρω ότι θα είναι πάντοτε ε, στην ακρόασή μας. Ο κύριος Λαβία ε, με βοηθάει να μαθαίνω τα Ιταλικά μου σιγά σιγά και έτσι Τζοβάνι σε διαβεβαιώ ότι στο τέλος του χρόνου θα τα έχω μάθει φαρσί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέραν των αστείων, έχουμε να κάνουμε μια περίοδο σχετικά δύσκολη, δηλαδή στο τέλο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα έχουμε πολύ στενά δημοσιονομικά περιθώρια, το είπε και ο εισηγητή. Και η κατάσταση ξέρουμε ότι θα είναι λιγότερο σοβαρή ενδεχομένω στην γεωργία, διότι υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερο από ότι σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό θα ήταν να μην ξεπερνούμε τα ε, ανώτατα όρια. Εάν επαναφέρουμε λοιπόν το προσχέδιο του προπολογισμού, νομίζω ότι το περιθώριο που θα έχουμε για επιπλέον προτεραιότητες θα είναι πάρα πολύ στενό. Ω εκ τούτου, για φέτο ή για τον προπολογισμό του 2013 καλύτερα, θα πρέπει να ορίσουμε και άλλε προτεραιότητε, ώστε, όπω είπε και ο Γενικό Συγητή, να είμαστε σε θέση εκεί όπου κάποιες γραμμές του προϋπολογισμού διαπιστώνεται ότι δεν αποδίδουν ή δεν απορροφούνται επαρκώς, να αξιοποιήσουμε το περιθώριο αυτών ή αν τα καταφέρουμε να έχουμε κάποιες επιπλέον προτεραιότητες, θετικές προτεραιότητες σε σχέση με την ε, δυνατότητα να αξιοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια ή αρνητικέ προτεραιότητε σε περίπτωση που δεν φτάνουν τα κονδύλια. Και αυτό γιατί βέβαια δεν ε, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πάντα πλεονάσματα και ίσω θα πρέπει να αναζητούμε και από πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων. Εφόσον λοιπόν τα κράτη-μέλη έχουν βάλει πλώρη για λιτότητα, για προπολογισμού λιτότητα, πρέπει και εμεί αντίστοιχα να επιδείξουμε πνεύμα υπευθυνότητα. Για τα πιλωτικά προγράμματα, για τα προγράμματα δράση που αναφέρθηκαν και τα δύο ζητήματα είναι πολύ σημαντικά για τη γεωργική πολιτική. Καταρχά, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι προτεραιότητέ μα και προφανώ έχουμε σε πιθανότητες επιτυχίας ε, ως προς τις προτάσεις μας Επιτροπής των Προπολογισμών εφόσον είναι οι προτάσεις αυτές ε, λογικές και ε, κοινέ μεταξύ διαφορών ομάδων, δηλαδή όχι χωριστά και αποκομμένα προγράμματα ή έργα. Επίση, στι προπαρασκευαστικέ δράσει και τα πιλωτικά προγράμματα, σημαντικά μου φαίνεται ότι εάν μπορέσουμε να επιτύχουμε και να πείσουμε του συναδέλφου μα από την Επιτροπή των Προπολογισμών ότι έχει σημασία ιδιαίτερη κάποια δράση, ένα πρόγραμμα, όταν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Προπολογισμών αποφασίσουν να το χρηματοδοτήσουν το εν λόγω έργο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανασκουμποθεί και εκείνη και να υλοποιήσει τι προτεραιότητε που θα έχουμε εμεί προσδιορίσει. Πολλά από τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία σε προηγούμενα έτη είχαμε χαρακτηρίσει χαρακτηρίσω σημαντικά και κοιτάω και στο, και προς τον κύριο Μποβέ γιατί εκείνος είχε ε, διατυπώσει την έκθεση για την αλυσίδα των τροφίμων και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτήν και ως αποτέλεσμα αυτής της εκθέσεως κύριε Μποβέ κάθε χρόνο δούμε ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας για να καταγράφονται οι τιμές και οι εξελίξεις στις τιμές. Η ΔΕ Επιτροπή μας είπε, α, ευχαριστούμε πάρα πολύ Επιτροπή της Γεωργίας, ένα εκατομμύριο σε δυσμένες υποχρεώσεων και 500.000 ευρώ σε πληρωμές μας δώσατε μεν, εμείς όμως θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερε πληροφορίε. Εμεί έχουμε αρκετέ πληροφορίε στη θέση μα. Ε, και εγώ απαντώ, εν πάση περιπτώσει, αφού έχετε αρκετέ πληροφορίε, τότε να μα τι κοινοποιήσετε και εμά, γιατί δεν αρκεί να καταλήγετε σε συμπεράσματα, πρέπει και αυτά τα συμπεράσματα να κοινοποιούνται, να είναι γνωστά και σε άλλου. Αυτό λοιπόν και θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να καλέσουμε την Επιτροπή Προέδρε, αν όχι σήμερα πάντω σε μια άλλη ευκαιρία, να μα εξηγήσει γιατί ορισμένε από τι προτεραιότητέ μα δεν υλοποιούνται. Μια από τις, ε, κάποιες από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να προσδιορίσουμε ως Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να προσδιοριστούν από κοινού, όπως είπα νωρίτερα, δηλαδή τιμές, περιθώρια, ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί στον προπολογισμό για το επόμενο έτος θα είναι η κατάσταση των χώρων των απορροκυπευτικών, των κυπευτικών καλύτερα. Ε, είχαμε τη μεγάλη κρίση που διαθέσαμε από τον τρέχοντα προπολογισμό Κονδύνα και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη περιμένει τη συγκεκριμένη πρόταση για να ε, απελευθερώσει τα κονδύλια, άρα περιμένουμε αυτό και επίσης στρεφόμενοι και προς την Esther Rans, ε, ε, λέω ότι εργάστηκαμε, εργάστηκε με ε, αντίξωες συνθήκες στον τομέα αυτό και Ίσως η πρόθεση των, προϊόντων αποτελεί μια καλή λύση. Κοιτάω και τους άλλους και τους για να δω τι άποψη μπορεί να έχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτά. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ τον Γενικό Εισηγητή. Περιμένω να ακούσω και τους λοιπούς ε, συναδέλφους και οδησηγητές και θα τα πούμε μετά. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, είχαμε την ευκαιρία να είναι εδώ ο συνάδελφος Ζωβάνη Λαβία και, που είναι και γενικός συγητής και άρα να δώσουμε μεγαλύτερη βάρος στον ρόλο της Επιτροπής μας. Πρώτα ο Τζόρτζο Λάιον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προσέγγιση της Έστερ για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ετοιμάσει τις προτεραιότητές της η Γεωργική Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας μας, είναι κάτι πολύ σωστό. Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα δηλαδή και πώς θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία της Επιτροπής μας. Αυτό θα φανεί από τις προτάσεις που θα κάνουμε για τον προπολογισμό. Όντως, θα περιοριστούν πολύ τα χρήματα και ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη ζητούν ε, χρήματα για να αντιμετωπίσουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς με τις προτάσεις μας θα καταφέρουμε παρόλα αυτά να ε, εξοικονομήσουμε χρήματα. Προτεραιότητά μας βέβαια είναι ο γεωργικός προπολογισμό. Δεύτερον, τα πειραματικά προγράμματα. Ναι, Ελπίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία τελικά μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων για να το υποστηρίξουμε αυτό. Εγώ θα προσπαθήσω να το πετύχω, να συζητήσω με τους άλλους σκιώδεις, ώστε να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική διαπραγμάτευση αυτή που θα κάνουμε για τον προπολογισμό του 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, George και ο Τζόρτζ είναι σημαντικός, ε, παίζει σημαντικό ρόλο γιατί είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον προπολογισμό του 2013, έστω και αν η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι διαθέσιμη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Εστέρ, τον Τζοβάνι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί. Επίσης, ε, σαφές είναι ότι ο προπολισμό του 2013 λόγω των άδειων ταμείων και των μεγάλων περικοπών στα κράτη-μέλη υφίσταται σημαντικές πιέσεις. Με δεδομένο αυτό, λοιπόν, θα ήθελα για άλλη μια φορά να επισημάνω πόσο μεγάλη σημασία θα είχε το να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα τους ε, ιδίους πόρους δεδομένης ε, της ε, στενότητας στο, στα δημοσιονομικά περιθώρια, καλό θα ήταν να προσδορίσουμε πολύ επακριβή ε, μέτρα και γι' αυτό καλό όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας με σοβαρότητα να αναλογιστούν ποιοι είναι οι τομείς εκείνη του προπολογισμού του 2013 που θεωρούν πιο σημαντικούς από τους άλλους. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, πιστεύω ότι σκόπιμο θα ήταν στην Επιτροπή Γεωργίας να επικεντρωθούμε σε δύο ή τρία πιλωτικά προγράμματα στα οποία θα συμφωνήσουμε, στα τα οποία θα κρίνουμε όλοι ε, ενδιαφέροντα, σημαντικά. Και βέβαια και το Συμβούλιο από πλευρά του θα πρέπει να προσδιορίσει προτεραιότητε και να εξηγήσει και τι περιμένει επακριβώ από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μεταφέρονται όλο και πιο πολλοί τομεί δραστηριοτήτων, αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεν, αλλά ο προπολογισμό τη διαρκώ να να συρρυκνώνεται. Δεν είμαστε πια, 20, δεν είμαστε πια 15 κρατημέρια, αλλά 27. Και ως το χρειαζόνται και τα σχετικά κονδύλια. Γιατί τη γεωργία χρειαζόμαστε έναν ε, προπολογισμό εύρωστο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην μόνο ποτέ ότι η γεωργική πολιτική είναι η μοναδική το όντι κοινοτικοποιημένη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό από αυτό θα εξαρτηθεί και η συνέπεια στους επιμέρους τομείς πολιτικής, γιατί δεν είναι δυνατόν, παραδείγματι, μέσω των επιδοτήσεων των εξαγωγών να προξενούμε αρνητικές ή αντίξωσες συνέπειες ε, στην παραγωγή μας. Γι' αυτό ε, χαίρομαι ιδιαίτερος, περιμένω μάλλον να ακούσω με αδημονία στις 25 Απριλίου τον προπολογισμό, την πρώτη προπολογισμού θα έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γέγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα όλα αυτά τα χρόνια για την Επιτροπή μας συζητάμε. Ευχαριστώ και τον Τζοβάνι και την Έστερ. Έχουμε, πιστεύω, μια καλή ομάδα που αγωνίζεται για τα θέματα αυτά και άρα μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητες. Πάντα γίνεται λόγος για λιτότητα για εξοικονομήσει πόρων. Και βεβαίω το σέβομαι αυτό. Βεβαίω δέχομαι ότι εφόσον επιβάλλεται η λιτότητα στου εθνικού προπολογισμού, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Αλλά κοιτώντα μόνο την περίπτωση τη την περίπτωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όταν έχουμε μόνο 1% από, την, ε, από το προϋπολογισμό μας που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έπρεπε τα ευρωπαϊκά κράτη, τα κράτη-μέλη δηλαδή, τα οποία βεβαίως και είναι υποχρεωμένα να κάνουν ε, ε τις οικονομίες τους, αυτό το πεδίο ε, αυτό το πεδίο ε, αυτή την αναλογία δηλαδή επί του προπολογισμού δεν θα πρέπει τουλάχιστον να τη λάβουν υπόψη και να τη χρηματοδοτήσουν ικανοποιητικά και να μην φορτώσουν όλη την ε, λιτότητα πάνω σε αυτό το μικρό, πολύ μικρό ποσοστό της, ε, του προπολογισμού που χορηγούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αποκομίζουν πάρα πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Έτσι λοιπόν θα θέλω να πω ότι θα πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσουμε, να μεριμνήσουμε ιδιαίτερω δε για τους νέους και για την για να μην φύγουν οι νέοι από την Υπεθρό, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε πολύ χειρότερα προβλήματα και πολύ μεγαλύτερο κόστος φυσικά. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική και ιδιαιτέρως με έμφαση στην Ήπεθρο. Πρέπει, και θα συμφωνήσω εδώ ρητά με την κυρία Ρόντουστ, Πρέπει να αναλογιστούμε συγκεκριμένα και να ορίσουμε προτεραιότητες, να πούμε τι είναι σημαντικό για μένα, τι είναι λιγότερο σημαντικό και ασφαλώς αυτό θα πρέπει με το πνεύμα ομοφωνίας να το συστήσουμε στην ομάδα μας, στην επιτροπή μας και να ορίσουμε ώστε να μπορούμε να μιλάμε και με μία φωνή για το ποιε είναι οι προτεραιότητες για τη γεωργία στο επόμενο διάστημα. Ο γεωργικός προπολογισμό λοιπόν πρέπει για άλλη μία φορά να υπογραμμιστεί ότι εκφράζει τη μόνη κοινοτικοποιημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρος Ικέρης και μετά ο Γιάννη. Βιάστηκα, πρόεδρε, βιάστηκα, συγγνώμη. Ο κύριος Σικίωσκη. Ευχαριστώ. Αναφερθήκανε, αναφέρθηκε η εξοικονόμηση στον προπολογισμό. Σε τι κλίμακα όμως. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για τα διευθυντικά ταμεία κυρίως και όχι για την κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που πηγαίνει στα κράτη-μέλη είναι πόροι αναπτυξιακοί οι οποίοι μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Οπότε, πού θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, από πού. Και έπειτα Ποιο είναι το επίπεδο πόρων για το οποίο μιλάμε. Εξοικονομήσεις ε, δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Ρωτάω γιατί αν συμβεί να μην έχουμε να μην εγκριθούν οι δημοσιονομικές προπτικές, τότε το 2013 θα είναι μια σημαντική χρονιά σε σχέση με τα επόμενα χρόνια. Έχετε εκτιμήσει λοιπόν μήπως ποια θα είναι η αναλογία του γεωργικού προπολογισμού στο συνολικό προπολογισμό για το 2013 και για την εφταετή περίοδο. Γιατί αν έχουμε την έκφραση αυτού του ποσοστού, τότε θα ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι η μείωση για την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ κύριο Γιώργ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω μερικέ παρατηρήσει και εγώ. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστώ του δύο συγκητέ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο γεωργικό προπολογισμό και από του δύο ε, και στο πρόσωπο μάλλον των δύο συγκητών έχει βρει αντάξιους υποστηρικτές Και ε, ξέρουμε βέβαια ότι καλό θα είναι τα στρατεύματα του ίδιου στρατηγού να μην ε, βρίσκονται σε αντιπαλότητα μεταξύ του, δηλαδή να συνεργάζονται και να τίνουν προ τον ίδιο στόχο, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λιτότητα. Λιτότητα παντού γίνεται λόγο για τη λιτότητα και βέβαια προφανώ δεν θα είναι καθόλου καλό το να ακουστεί ότι εμεί στι χώρε μα, να ακουστεί στι χώρε ότι γίνονται, ε, επιβάλλονται μέτρα λιτότητα και γίνονται αιματηρέ ε, οικονομίε, αλλά αυτοί στι Βρυξέλλε δίνουν όλο και πιο πολλά ε, χρήματα για τον προπολογισμό του. Πολύ καλά όλα αυτά. Πλην όμω και εγώ Ενοχλούμε βαθύτατα από τα κράτη-μέλη τα οποία ζητούν όλο και πιο πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όμως να την καλύπτουν και οικονομικά. Ε, με την απαραίτητη χρηματοδότηση. Δηλαδή, όλο και πιο πολλά πράγματα συστούμε για τι αρμοδιότητε Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, όμω χωρί καμία επάρκεια στην ε, χρηματοδότηση. Είτε πρόκειται για μεγάλα έργα, είτε πρόκειται για άλλα πράγματα. Ε, όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναλαμβάνει να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Τρίτη παρατήρηση. Γεωργικό προπολογισμό, και συμφωνώ εδώ με του προλαλήσαντε. Έχουμε νομίζω να επιδείξουμε τα τελευταία χρόνια μια καλή και λογική πολιτική. 17,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, στον πρωτογενή τομέα μόνο και προφανώς ε, ακόμη περισσότερες και στους συναφείς τομείς. Ε, κοινοτική δράση, κοινοτική πολιτική. Και πρέπει να πω ότι λυπούμε και εκνευρίζομαι βαθύτατα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αντιληφθεί το, με πόση σοβαρότητα συζητούμε τις ε, γεωργικές δαπάνες και πάντα προσπαθούν να παρουσιάσουν τα πράγματα διωγγωμένα γιατί εμείς εδώ προσπαθούμε όντως και κάνουμε πάρα πολύ προσεκτική δουλειά και επιλέγουμε τα σημεία στα οποία όντως χρειάζεται και να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας και να προστατέψουμε την ύπεθρο δεύτερο πυλώνα που ακούστηκε και νωρίτερα ε, και να έχουμε τα μέτσα εκείνα τα οποία θα στηρίξουν την ε, οικονομία στην ύπεθρο με πάρα πολύ λογικό τρόπο. Και θα ήθελα να επισημάνω επίση μια προτεραιότητα την οποία θα ήθελα εγώ να ζητήσω στον προπολογισμό, δηλαδή για τη γεωργία. Θα ήθελα να δω επαρκή ευελιξία. Δεν θα μίλησω για αποθεματικά, γιατί αυτό πιο πολύ μας παραπέμπει σε λογιστικά βιβλία. Αλλά θα ήθελα να υπάρχει μια ευελιξία έτσι ώστε εάν υπάρχουν κάποια μέτρα για την οργάνωση της αγοράς, εάν προκύψει κάποια φυσική καταστροφή, εάν χρειαστεί δηλαδή να κινητοποιηθεί ο γεωργικός προπολογισμό για να χρηματοδοτήσει κάτι το έκτακτο, για να μην χρειάζεται να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη επιπλέον χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο θα μα οδηγήσει βέβαια σε απώλεια σημαντικού χρόνου, θα ήθελα να έχουμε την ευελιξία να αντλήσουμε μέσω στα κονδύλια εκεί όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ, Σμιτ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί διάφορα ήδη υπόθηκαν και επίση ε, συμφωνώ με την προσέγγιση τη εισηγήτρια. Η Επιτροπή μα πρέπει να είναι ρεαλιστική και είναι αποκαλυπτική για το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις συζητήσεις για το πολιετές ε, πλαίσιο. Επίση μου άρεσε τα όσα είπε η κυρία Ντελάνγκη γιατί όλα είναι προτεραιότητα και τίποτα δεν είναι προτεραιότητα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί όμως για το πού θα κάνουμε οικονομίες και πού θα δαπανηθούν τα, τα χρήματα. Εμείς στο κοινοβούλιο κάνουμε λες και είμαστε παιδάκια και φτιάχνουμε το γράμμα στον Αϊ Βασίλη για, με τις επιθυμίες μας. Συνήθως. Ε, η ομάδα μας επίσης ε, πρότεινε την, ε, την δημιουργία του παρατηρητηρίου για τις τιμές και τα περιθώρια και εγκρίθηκε η πρόταση αυτή για να μπορούμε καλύτερα να αξιολογήσουμε τα όσα γίνονται στην αγορά. Τελικά βέβαια μέχρι να φτάσει στην Κομισιόν ε, μετατράπηκε σε υποσημείωση αυτό το αίτημά μας και ακόμα δεν έχουμε τα σχετικά στοιχεία. Αν υπάρχει λοιπόν η αίσθηση στην Επιτροπή ότι δεν ε, χρειάζεται να το κάνουμε, εντάξει, να μην το κάνουμε. Αλλά από τη στιγμή που εμεί θέλουμε προτεραιότητε, εμεί είμαστε οι δημοκρατικά εκλεγμένοι νομοθέτε, αναμένουμε να εφαρμοστούν όλα αυτά. Μια υγιή συζήτηση λοιπόν για το πού ακριβώς, ποιες ακριβώς είναι οι προτεραιότητες μας και τι συμβαίνει σε αυτές. Εγώ μένα μου αρέσει ο τόνος της συζήτησης λοιπόν και θα σας υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, κυρίως τους εισηγητές. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον ε, κύριο Λόγκο και μετά στην Ντελάγκη και στον Λαβία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια σύντομα σχόλια για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία παρακολουθήσαμε σήμερα το πρωί. ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του κυρίου Λαβία και τον, για τις κατευθυντήριες γραμμές που κατ' ουσία μας βρίσκουν σύμφωνους. Θα πρέπει ωστόσο να βρεθεί εδώ μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απέτηση για λιτότητα, στη προϋπολογισμό και μια άλλη επιτακτική ανάγκη, την οικονομική ανάκαμψη. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτές τις πτυχές και κυρίως την οικονομική ανάπτυξη στις ε, γεωργικές περιοχές που, όπου όπως τονίστηκε υπάρχει αυτή η ευαισθησία, αυτός ευάλωτος χαρακτήρας και χρειάζεται να υποστηριχθούν οι περιοχές της ε, υπαίθρου και δεν μπορεί η οικονομία των γεωργικών περιοχών να αντέξει μια ενδεχόμενη διακοπή της στήριξης. Όπως είπαμε, οι υπηρεσίε της Επιτροπής ε, προετοιμάζουν την πρόταση προπολογισμού για το 2013 για να θα εγκριθεί στι 25 Απριλίου και έλεγα και επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά ότι δουλεύουμε επί τη βάση συγκεκριμένων σενάριων που είναι συνεκτικά και σε συμφωνία με τις προβλέψεις του κυρίου Λαβία και που συμφωνούν με τα όσα σύστησε και η κυρία Ντελάγκε στη διάρκεια της παρέμβασης της. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία προϋπολογισμού είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ότι είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός των συγκεκριμένων δημοσιονομικών προοπτικών και εν είναι δύσκολη, η, δύσκολο το εγχείρημα λόγω των οικονομικών περιστάσεων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση λείπει μια ερώτηση, ε, δεν έγινε μια ερώτηση, την οποία είχα προετοιμαστεί να απαντήσω και πιστεύω πως είναι μια ανησυχία που σε αυτή την περίοδο του χρόνου εμ, απασχολεί όλους όσου ασχολούνται με τη γεωργία και είναι το κατά πόσο θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Χωρίς να θέλω να προτρέξω τις προθεσμίες της 31ης Μαρτίου, μπορώ να σας πω πως υπάρχει κάποια ηρεμία στην ε, Κομισιόν όσον αφορά το συγκεκριμένο ρίσκο. Δεν θα πρέπει να επιβληθεί η δημοσιονομική πειθαρχία φέτος, και χάρη και στο γεγονός ότι Υπάρχει ένα υπόλοιπο στο Ταμείο Αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης της τάξης των 640 εκατομμυρίων ευρώ. Πράγμα από το οποίο θα μας ε, βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ε, δημοσιονομική πειθαρχία φέτος. Αυτό είναι καλό νέο λοιπόν, αλλά είναι και μια ανησυχία που θα ήθελα να τονίσω, δηλαδή το γεγονός ότι όπως υπόθηκε βρισκόμαστε σε μια προηγμένη φάση του προγραμματισμού για τα προγράμματα ε, τη... τα πολιετή που θα επιταχυνθεί η φάση αυτή λόγω της εφαρμογή και της ολοκλήρωσης αυτών των προγραμμάτων και γι' αυτό και θα υπάρξει μεγαλύτερη απέτηση όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και από αυτή την άποψη ελπίζω πως από πλευράς της Επιτροπής Γεωργίας και των εισηγητών Λαβία και Ντελάγκε θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την πτυχή που μας ανησυχεί. Όσον αφορά εμένα λοιπόν, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόγκο και σας ευχαριστούμε και για τα νέα αυτά που μας δώσατε. Και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Ντελάγκη και αν χρειάζεται και τον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ πολύ, θα σύντομη. θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. για τις ε, προτεραιότητες, τα θέματα τα οποία θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά και που έθιξαν στις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που ήρθε με τον εκπροσωπό της που, μας, ε, ε, που συνεργάζεται μαζί μας. Και θα ήθελα επίσης ιδιαίτερος να αναφερθώ στα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις πολύ σημαντικό παράγοντα και είναι σημαντικό να γίνει η συζήτηση αυτή εις βάθος όχι μόνο για τις ε, προτεραιότητες ε, που έχουμε για το μέλλον, αλλά και για τις προτεραιότητες που εύλογα είχαμε προσδιορίσει και στο παρελθόν. Και καλό θα ήταν να δούμε, εάν υπάρχει δυνατότητα βέβαια, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο, ο οποίο θα μα εξηγήσει γιατί Φερρυπίν στο περιθώριο για τις μάλλον στο παρατηρητήριο για τα περιθώρια και τις τιμές, δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Και επίση άλλον, νομίζω ότι στρεφόμενοι προς όλες τις πολιτικές ομάδες μπορώ να διαπιστώσω ότι ο κάθε ένας μας, η κάθε πολιτική ομάδα έχει κατά καιρού ε, στηρίξει το αίτημα αυτό και προβάλλει το αίτημα αυτό. Μπορεί μεν να το σημειώσαμε ξεκάθαρα στην έκθεση Μποβέ, αλλά και το ΕΡΚ και οι σοσιαλιστές έχουν κατά καιρού τοποθετηθεί στην υπόθεση αυτή. Εν πάση περιπτώσει αφορά εμάς, ε, ιδιαίτερα θέλουμε να δούμε τι ε, αποδοτικότητα έχουν προγράμματα, έργα τα οποία έχουν αρχίσει να λειτουργούν και τι, τι κάνει με, σε σχέση με αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, περιμένω να τις ακούσω. Τζοβάνι. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους για την ενδιαφέρουσα συζήτηση για την δυνατότητα που μου δώσατε να ακούσω σύντομα, ε, χρήσιμες συμβολές για τις εργασίες που θα κάνουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις που νομίζω θα είναι χρήσιμες. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, θα πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι τα περιθώρια που έχουμε διαθέσιμα στους διάφορους τίτλους και δεδομένη της δυσκολία των κρατών μελών θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διαθέσουμε στους ε, εκάστοτε τίτλους και κατηγορίες συγγνώμη και επίσης ε, να απαντήσω και στον Πίτερ Γιάρα που αναφέρθηκε στην απαραίτητα ευελιξία για τις ε, παρεμβάσεις κρίσης. Όπως όλοι γνωρίζετε, στο εσωτερικό του ε, προπολογισμού έχουμε την, την ανάγκη και την υποχρέωση να διατηρήσουμε ένα περιθώριο 300 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις επίγουσας ανάγκες και πιθανότατα αυτό θα συνεχιστεί και για τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Δεμό όμως, τον προπολογισμό του 2013 σίγουρα θα διατηρήσουμε το υποχρεωτικό περιθώριο. Αντί ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι επειδή είναι το τελευταίο έτος της, του πολιετούς πλαισίου, δημοσιονομικού πλαισίου, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο προπολογισμό του 2013 θα μπορούσε να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα διοργανική συμφωνία θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο προπολογισμό να θεωρηθεί ως βάση για ε, ενδεχόμενη εκτέλεση του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιο αν δεν υπάρξει συμφωνία ή ομοφωνία εντός του Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το προπολογισμού του 2013 θα χρησιμοποιηθεί ως βάση με την προσθήκη βέβαια του πληθωρισμού. Τελευταίο στοιχείο αφορά τις προτεραιότητες. Τις τελευταίες δύο δημοσιονομικές διαδικασίες τις οποίες παρακολούθησα στο πλαίσιο της Επιτροπής Προπολογισμού και στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής είδαμε πως τελικά το Συμβούλιο ήρθε στην ε, συνδιαλλαγή με περιορισμένη διαθεσιμότητα όσον αφορά τα κονδύλια για τις πιστώσεις πληρωμών με συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένα όρια χωρίς να υποδεικνύει πού θα πρέπει να γίνουν οι περικοπές και αυτό εμείς το τονίσαμε ε, στις μα μας γραμμές και είπαμε ότι όταν θα θέλει το Συμβούλιο να μας δείξει συγκεκριμένες προτάσεις για μικρότερη αύξηση από αυτή που προτείνει η Κομισιόν και με βάση τις δικές εκτιμήσεις θα πρέπει να μας πει και πού θα πρέπει να κάνουμε κάνουμε τις περικοπές. Να μην μας αφήνει εμά δηλαδή την ευθύνη για τις εν λόγω περικοπές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί και η σύγκριση που μπορώ να κάνω με όλες τις άλλες περιτροπές που γερνάω εδώ στην ε, δικιά σας θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι εδώ γίνεται δουλειά, γίνεται δουλειά συγκεκριμένη και η συμβολή σας στη συζήτηση αυτό δείχνει. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε τακτικά. Θα τα λέμε μάλλον τακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε κύριε Λαβία και θα συνεχίσουμε με αυτό το τόσο κρίσιμο σημείο. Και περνάμε στο επόμενο στην ημερήσια διάταξη. Ο Nicholson. James Nicholson είναι εδώ και θα εξετάσουμε μαζί ε, το 10 και το 11 που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 64432 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη-μέλη. Και το επόμενο θέμα που είναι το 11 αφορά την προαιρετική επισήμανση του βοήου κρέατος και θα τα εξετάσουμε από κοινού. Ο εισηγητής είναι ο ίδιος, ο Τζιμ Νίκολσον, του δίνω το λόγο και είναι παρόντες διάφοροι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και για τις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις είναι στη 29η Μαρτίου. Λίγες μέρες έχουμε ακόμα δηλαδή. Έχεις Τζιμ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, είναι δικιά μου, δικό μου θέμα αυτό. Το ανέλαβα από την Επιτροπή και πρόκειται για την πρόταση της ε, Επιτροπής όσον αφορά ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων ε, επιτήρησης και για διαγραφή των διατάξεων ε, σχετικά με προαιρετική επισήμανση. Όντω υπάρχουν ε, ηλεκτρονικές ε, βάσεις δεδομένων στα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ε, πω λιγάκι τι έχω κάνει όσον αφορά την ταυτοποίηση των βοηδών και μετά για την σήμανση. Το, ο βασικός στόχος είναι να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων και να αποτελεί αυτό το πιο βασικό τρόπο για να αναγνωρίζονται τα ζώα αυτά. Λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχει ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Η πρόταση επίσης έχει ως στόχο να εισαγάγει εναρμονισμένες υψηλές προδιαγραφές έτσι ώστε να έχουμε την βέλτιστη ηλεκτρονική αναγνώριση και να υποφεληθούμε από όλα τα τεχνικά πρότυπα. Το ότι μιλάμε για θελοντική βάση ή για το ότι κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν ε, να είναι υποχρεωτική εθελοντική αποτελεί και αυτό ε, μέρος της προσέγγισής μας γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υποφεληθούν οι γεωργοί από την ε, τεχνολογία μπορούν να το κάνουν εφόσον θέλουν ενώ άλλοι μικροί ίσως γεωργοί που δεν έχουν να από αυτό μπορούν να επιλέξουν να μην το κάνουν. Στηρίζω την προσέγγιση αυτή, όμως έχω υποβάλει και μία ε, τροπολογία η οποία ε, προβλέπει μία εξαίρεση. Και μιλάμε για δύο είδη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τώρα όσον αφορά για την διαγραφή των ε, διατάξεων σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοήου κρέατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν οι διατάξεις αυτής. Έχουμε παραδείγματα τέτοιας ε, σήμανσης στα σούπερ μάρκετ ε, και σε άλλα καταστήματα. Με το τρέχον σύστημα οι φορείς έπρεπε να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κράτους μέλους τους προτού να μπορέσουν την σήμανση αυτή να την βάλουν στο πακέτο. Όμως η διαδικασία αυτή, από ό,τι φαίνεται, έγινε υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος χωρίς να προσφέρει καμία προστιθόμενη αξία στον καταναλωτή. Δεν υπήρχε τίποτα που να το δικαιολογεί δηλαδή πια. Οπότε χαίρομαι που ε, υπάρχει η διαγραφή αυτή γιατί έτσι απλοποιούμε τις διαδικασίες. Ο καταναλωτής μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι δεν πρόκειται για μείωση των προδιαγραφών και ότι η ασφάλειά του καλύπτεται πλήρως και έχει τις πληροφορίες που πρέπει. Κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να πούμε πριν από λίγο καιρό. Στηρίζουμε λοιπόν την ε, πρόταση αυτή και τη στηρίζει και η Επιτροπή ΕΝΒΗ. Τώρα όσον αφορά την εποπτεία στα κράτη-μέλη, εδώ πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπληρώνει τις δικές μου προτάσεις. Το συζήτησα λίγο για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ε, ταυτότητας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση των βοηδών. Και από ό,τι φαίνεται, τα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη ανταποκρίνοντας τις προδιαγραφές. Θα ήθελα όμως εδώ πέρα να προσθέσω κάτι όσον αφορά την χρήση της ηλεκτρονικής αυτής ταυτότητας. Δεν έχω υποβάλει μένα τροπολογίες στην πρόταση αυτή, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η άποψη των γεωργών γι' αυτό. το θέμα της τιμής της τεχνολογίας. Σίγουρα η τιμή θα μειωθεί και έτσι θα είναι πιο ελκυστική επιλογή. Σίγουρα θα διευκολύνει τη ζωή των ε, γεωργών. Θα ξέρουμε θα είναι πιο εύκολη η χνηλασιμότητα, η διαχείριση των ε, κοπαδιών τους. Οπότε με τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα στο μέλλον αυτό θα αποτελέσει κάτι πολύ σημαντικό για τις εξαγωγές μας προς άλλες χώρες που τα χρησιμοποιούν ήδη αυτά τα συστήματα. Αλλά είναι καλό το ότι είναι σε θεωρητική βάση ακόμα. Ίσως ε, κάτι έμαθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από άλλα επίμαχα αντίστοιχα θέματα που είχαμε. Οπότε ευτυχώς το βάζει σε θελοντική βάση αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ε, πληροφορίες αυτές που μας δώσατε και για την εισαγωγή που κάνατε. Η κυρία Γκαρσία Πέρες έχει ζητήσει το λόγο και μετά κύριε Ράιμερς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Νίκολσον για τα όσα μας είπε. Θέλω και εγώ να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που έθεσε και εκείνο. Πρώτον, να πω ότι συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής και εμείς για την διαγραφή της ε, θελοντικής ε, προαιρετικής επισήμανσης του βοηού κρέατος. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι από τη στιγμή που άρχισε προαιρετική επισήμανση έχει τροποποιηθεί η αγορά βοηού και πρέπει να αναθεωρηθεί το υπάρχον σύστημα. Όμω πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, το σύστημα αυτό ήταν ε, αποτελεσματικό μέχρι που άρχισε να ζητάει τη ρύθμιση του ο κλάδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να γίνει αναθεώρηση, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε το διοικητικό άχθο να είναι παραπάνω από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος αυτού, γιατί αλλιώς δεν θα το ήθελε ο κλάδος. Για μας η ρύθμιση μέσω των οριζοντίων υπαρχουσών διατάξεων είναι κάτι που φτάνει χωρίς να είναι πολύ φιλόδοξο και αυτό και προτείνουμε κάτι να γίνει κάθετα ανάλογο όπως έχουμε με τα, τα πτηνά για παράδειγμα. Αυτή η κάθετη προσέγγιση θα έχει γενικό χαρακτήρα και υπάρχει στον, ε, στην ενιαία οργάνωση αγοράς και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναφέρεται ο κανονισμός αυτός όπως επίσης και άλλα οριζόντια μέτρα. Όπως και να έχει το πράγμα πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κινητικό πλαίσιο για την προαιρετική επισήμανση του βοήου κρέατος όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς, τα πτηνά για παράδειγμα ή άλλα είδη κρέατος. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρχει αναρμόνιση μέσα στην ενιαία αγορά χωρίς να έχουμε στρεβλώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Ράμες και με τα κυρία Κώσταγκερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. η σημασία έχει βέβαια η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον κανονισμό. Θα ήθελα ωστόσο να καταστήσω και σαφές ότι ιδιαίτερα η ηλεκτρονική επισήμανση βοηδών με ενδιαφέρει. διότι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ύστερα από τόσα χρόνια που λειτουργεί ότι είναι ε, απρόσκοπτη η λειτουργία αυτού του συστήματος ηλεκτρονικής επισήμανσης. Βλέπουμε ότι σε περίπτωση ελέγχων, εάν το ηλεκτρονικό σύστημα για κάποιο λόγο παραδώσει το πνεύμα ή δεν λειτουργεί σωστά, δεν έχει τη δυνατότητα ο Γιώργος να αποκαταστήσει και να εξηγήσει ότι το πρόβλημα ήταν μόνο τεχνικό και να δείξει ότι έχει κάνει σωστή επισήμανση. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο επίπεδο αυτό και ένα ηλεκτρονικό ε, ένα ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα μια γεωργική εκμετάλλευση. Άρα καλό θα, έπρεπε, θα ήταν πιστεύω να εισαγάγουμε και ένα περιθώριο ανοχής στα συστήματα αυτά. Ναι, να εισάγουμε λοιπόν τα σύγχρονα συστήματα, τη νέα τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε με, μια, με ένα βαθμό ευελιξίας και το περιθώριο να εξοικειωθεί ο χρήστης με τα συστήματα αυτά, αλλά και να αποδεχθεί την τεχνολογία αυτή και μόνο όταν θα είναι αποδεδειγμένα χαμηλό το ποσοστό σφάλματος να εισαγάγουμε με πιο αυστηρούς όρους, να ορίσουμε πιο αυστηρούς όρους για τη τεχνολογία αυτή. Διότι, επαναλαμβάνω, αν το κάνουμε με τη βία, ε, αν επιβάλλουν τα κράτη-μέλη άνωθεν αυτούς τους, ε, αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα και αντίσταση στεναρή από ε, τους ε, κτηνοτρόφους. θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν είχαμε τα παραδοσιακά ενότια, είναι πολύ απλό ο έλεγχο να πάει κάποιο μέσα στο στάβλο να κοιτάξει αν το ζώο έχει το ενότιο και να διαπιστώσει την τήρηση των διατάξεων περί επισήμανση. Όταν όμω έχουμε το σύστημα το ηλεκτρονικό, πρέπει ο, καθένας να περνάει, πρέπει ο ελεγκτής να περνάει με ένα σκάνερ από το κάθε ζώο για να, δια, για να βεβαιωθεί καταρχά εάν δουλεύει το μηχάνημα, αν εκπέμπει δηλαδή το, το τσιπ. Και γι' αυτό ε, καλό θα ήταν τα μέτρα που εισάγονται και να γίνονται ε, να εισάγονται σε πνεύμα συζήτησης ε, θελοντικό ενδεχομένως, ώστε να υπάρχει επαρκής αποδοχή από τον Γεωργό, να τον πείσουμε ότι ε, το σύστημα αυτό είναι προς όφελός του και προς συμφέρον του. Και ότι, λειτουργεί σωστά. Ευχαριστούμε. Κέστιγκερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τον Τζέιμς Νίκολσον που ανέλαβε να εκπονήσει την έκθεση για το θέμα αυτό. Εμεί, ε, εκπροσωπώντα τον κόσμο τη Γεωργία, προφανώ και έχουμε κάθε ενδιαφέρον να είναι εφαρμόσιμα στην πράξη τα μέτρα που προτείνονται και βέβαια η τεχνολογία στα συστήματα επισήμανσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προόδου. Εγώ προσωπικώς είμαι κατά της διαγραφής των διατάξεων περί της εκούσιας επισήμανσης, ηλεκτρονικής επισήμανσης. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε εν γέννη εισαγάγει στην Αυστρία μέσα από τέσσερις διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη διάχυση των προϊόντων στην αγορά, το οποίο στηρίξαμε ακριβώς στο εκούσιο σύστημα επισήμανσης και ε, βλέπουμε ότι είχε μεγάλη επιτυχία, είχε επιτυχία και σε επίπεδο καταναλωτή ο οποίος ζητά τα προϊόντα, ζητεί τα προϊόντα αυτά και άρα μπορούμε να ε, πούμε ότι ήταν επιτυχημένο το σύστημα. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω με οποιαδήποτε πρόταση έχει να κάνει με περιστολή της γραφειοκρατίας, του διοικητικού φόρτου, διότι προκαλώ, προφανώς ε, αυτά παρεμποδίζουν ε, και την ε, δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής του συστήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η άρση της γραφειοκρατίας θα οδηγήσει σε ένα σύστημα αδιαφανές, ένα σύστημα χωρίς ελέγχους, το οποίο θα είναι πρόσφορο σε καταχρήσεις και καταστρατηγήσεις της νομοθεσίας. Συμφωνώ λοιπόν και με την προλαλήσασα ότι θα πρέπει το πιθανό τεχνολογικό σφάλμα, ελάττωμα να μην αποβαίνει εις βάρος του ε, γεωργού. Εφόσον δεν είναι πια, δεν είναι ακόμη μάλλον όριμη τεχνολογικά η μέθοδος αυτή της, ε, της ηλεκτρονικής επισήμανσης, δεν μπορούμε να φορτώνουμε όλα τα φταξίματα στον γεωργό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να στηρίξω όλο είπε η κυρία Ρήμες. Εκείνη είναι γεωργός και ξέρει για τι πράγμα μιλάει. Είναι εκείνη λογική αυτά που λέει. Ένα σύστημα το οποίο δεν είμαστε σίγουροι για το πόσο αξιόπιστο είναι, μας οδηγεί σίγουρα στην καταστροφή. Δεν μπορεί να το κάνουμε υποχρεωτικό αν δεν είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί, σίγουρα ένα σύστημα που λειτουργεί διαχειριστικά βοηθάει. Και οι γεωργοί, η μεγάλη παραγωγή ε, κτηνοτρόφια γελών, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσουν για να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις αγέλες τους. Αυτοί όμως θα ελέγχουν και θα βλέπουν κατά πόσο λειτουργεί το σύστημα ή όχι. Αν όλοι αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, ίσως τότε να έχει νόημα να το επιβάλλουμε, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε καθόλου κατά πόσο θα λειτουργεί, οπότε δεν έχει νόημα. Ευχαριστούμε. Δεν ε, ζητάει κανένας άλλος το λόγο, οπότε ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής παρακαλώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, όλους όσοι πήραν το λόγο στην ε, συνάντηση αυτή. Έχουμε σημειώσει όλα τους τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες ε, απαντήσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση και στη συνέχεια όσον αφορά την προαιρετική επισήμανση. Έχω εδώ και τους συναδέρφους οι οποίοι θα έχουν και αυτοί πράγματα να σας απαντήσουν. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, μερικές ε, διευκρινήσεις που θα έπρεπε να δώσω για την ηλεκτρονική αναγνώριση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά άκουσα σχόλια από ορισμένου εδώ που λένε ότι η προαιρετική προσέγγιση είναι καλύτερη και όχι υποχρεωτική και επίσης αναφέρθηκαν και στις ανάγκη για διάλογο από πάνω προς τα κάτω. Αναφέρθηκαν επίσης και σε θέματα που έχουν που λένε εντάξει δεν το είπανε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αλλά το χρησιμοποιούμε σαν πειραματόζωα τους γεωργούς δεδομένου ότι δεν ξέρουμε ακόμα η τεχνολογία αυτή πόσο έγκυρη θα είναι. Εδώ θέλω λοιπόν να κάνω κάποιες διευκρινήσεις πολύ απλά. Ο διάλογος ε, αυτός τον οποίο αναφέρθηκε ε, κάποιος υπάρχει ήδη, έχει ήδη ξεκινήσει. Και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να γνωρίζει τι προβλήματα ενδεχομένω υπάρχουν. Δεν θέλει να υπάρχει ε, έλλειψη διαβούλευσης. Γι' αυτό και ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα από τον Οκτώβριο οργανώσαμε μια συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να τους πούμε κοιτάξτε ορίστε θα έχουμε ε, μια συζήτηση ας τα πούμε μεταξύ μας πείτε κατά τη γνώμη σας ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία για αυτή τη δουλειά βασισμένη βέβαια στην εμπειρία που έχετε εσείς επί τόπου. Όπως σας είπα προσπαθώ να τα πω σύντομα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε τότε ήταν ότι η τεχνολογία που έχουμε τώρα, που είναι το RFID, που είναι βάση συχνότητας ταυτοποίηση, εντάξει τώρα χαμηλή συχνότητα, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ανταποκρίνεται ε, πολύ καλά στις ανάγκες που έχουν οι γεωργοί για τις αγέλες τους. Σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιείται ήδη, υπάρχουν και ερευνητικά εργαστήρια που λένε ότι ναι, είναι κατάλληλοι. Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν το εξή. Ότι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι έχουμε υψηλά ποσοστά εγκυρότητα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης, πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα ώστε το transponder να είναι καλό αυτό που κυκλοφορεί δηλαδή στην αγορά και ανταποκρίνεται τις ανάγκες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούγονται ανησυχίες από την εμπειρία που έχουν ορισμένοι με άλλα είδη ζών. Αλλά το διάλογο τον έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη. Έπειτα η Επιτροπή πριν προτείνει κάποια τεχνολογία δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί σαν πειραματόζωα τους γεωργούς για να δει κατόπιν κατά πόσο λειτουργεί αυτή η τεχνολογία ή όχι. Να ξέρετε ότι για, άλλα, για τα άλογα, για παράδειγμα, ε, για ε, πρόβατα κτλ. χρησιμοποιείται ήδη η ηλεκτρονική αναγνώριση. Δεν ξεκινάει εδώ. Θέλω τώρα να πω στη δικιά σας ακριβώς επιτροπή, την Επιτροπή Γεωργίας, ότι είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τον κλάδο αυτό στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Δεν θέλουμε έναν ανταγωνιστικό τομέα. Όντως, έχουμε τους καλύτερους παραγωγούς ε, ευοίου κρέατος ε, στον κόσμο, αλλά να ξέρετε ότι και άλλοι και στην Αυστραλία και στην Αμερική έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αναγνώριση. Άρα πρέπει να προβληματιστούμε για το πού θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω προφανώς, άρα και το δικό μας σύστημα ειχνηλασιμότητας πρέπει να το κάνουμε και πιο γρήγορο και πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι απάντησε έτσι όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση και εφόσον μου επιτρέπει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέρφους από την DG για την προαιρετική επισήμανση του βόηου κρέατος. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συμπληρώσω και εγώ κάτι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκολσον για τις ε, γνωμοδοτήσεις του. Εξήγηση της πρότασής μας είναι ότι το σύστημα της ε, υποχρεωτικής ή προαιρετικής ε, επισήμανσης απορρέει από την κρίση που είχαμε της εγκεφαλοπάθειας των βοηδών, που δεν υπάρχει πια. Τότε ξεκινήσαμε. Τώρα θα γίνεται με το βόλιο κρέας ό,τι γίνεται και με τα άλλα είδη κρέατος. Όπως γίνεται για τα πουλερικά κλπ. Έτσι και αλλιώς ε, υπήρξαν ε, επικρίσεις για την ρύθμιση αυτή, ακριβώς γιατί δεν έχει πια νόημα και γι' αυτό αποφασίσαμε ε, την διαγραφή των σχετικών διατάξεων. Βέβαια κάποιες χώρες είναι επιφυλακτικές, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα με τα οριζόντια μέτρα υπάρχει η ίδια κάλυψη. Θέλω επίσης να σας καθισχάσω και για το εξή. Κάποιος αναφέρθηκε στο τι γίνεται ε, με το κρέας των πτηνών. Εδώ μιλάμε για προαιρετικούς όρους, όπως είπε και ο κύριος Νίκολσον. Οπότε μιλάμε για δύο διαφορετικά συστήματα. Προτείνουμε λοιπόν να διαγραφούν οι διατάξει του κανονισμού για το βόηο κρέα, που σημαίνει ότι και το βόηο κρέα αντιμετωπίζεται εφ' εξή όσον αφορά σχισμού κτλ. με τον ίδιο οριζόντιο τρόπο όπω γίνεται και με τα άλλα είδη κρέατο. Ευχαριστούμε. Οπότε, ο εισηγητής τώρα. Παρακαλώ, James Nicholson. Εκτό μικροφώνου ο κύριος Νίκολσον, δεν τον ακούμε. Σίγουρα ήταν ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Βέβαια, αν τα συγκρίνουμε με άλλα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή μας, δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό που ξεσηκώνει τα πάθη. Υπάρχουν άλλα θέματα που έχουν αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικά. Πάντως, ευχαριστώ την Επιτροπή και τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο και περιμένω να δω αν έχουν τροπολογίες να υποβάλουν. Δεν έχω καμιά αφιβολία ότι αν κοιτάξουμε λίγο πίσω τι γινόταν πριν την κεφαλοπάθεια των βοηδών, θυμάμαι ότι δεν τους άρεσε καθόλου στους γεωργούς να έχουν τσίψη, να έχουν τέλος πάντων ε, τα στοιχεία έτσι όπως ε, τα έχουμε τώρα. Τώρα αντίθετα δεν καταλαβαίνουν ε, πώς αργήσαμε τόσο πολύ να έχουμε τέτοια συστήματα υγνελισιμότητας. Όσο περνάει ο καιρός και όσο βελτιώνεται η τεχνολογία και όσο γίνεται και πιο φτηνή, τότε ναι, βεβαίως και να προχωρήσουμε. Ασφαλώς δεν λέω αν αυτό θα γίνει αύριο ή μετά από πέντε χρόνια, αλλά σίγουρα θα συμβεί όταν βιομηχανία σε λογικές τιμές μας δώσει τα κατάλληλα μέσα, προφανώς και θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα πάμε μπροστά μακροπρόθεσμα. Αλλά δεν θα πρέπει να βιαστούμε, δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε ε, τα πράγματα, αλλά να έχουμε υπόψη μας τι βελτιώσεις πρέπει ακόμα να γίνουν και πώς πρέπει να προχωρήσουν οι δοκιμές ώστε να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί και καλά το σύστημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλους και ό,τι τροπολογίες έχετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Προθέσουμε για την καθοστροπολογία 29 Μαρτίου το μεσημέρι στις 12 και νομίζω ότι να θα έχει τώρα να κοιτάξουμε και σε ποιο βαθμό αλλαγές πιθανές στα συστήματα τα ηλεκτρονικά μπορεί να κοστίσουν ή τι είδους δαπάνη συνεπάγονται. Ενώ να συζητήσουμε το 2013 και μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρήσιμη είναι η συζήτηση και τώρα σας ευχαριστώ και περνώ στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ήρθε από το, το επόμενο κομμάτι τη συνεδρίας, το απογευματινό δηλαδή, ένα θέμα το οποίο συχνά μας απασχολεί και που αφορά τις συνθήκες και την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά. Το λόγο θα λάβει τώρα ο εισηγητής κύριος Βορσισιόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έχετε λάβει, φαντάζομαι, το σχέδιο εκθέσεως μου για το θέμα αυτό. Το κείμενο που ετοίμασα σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές, ο οποίος και ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ανακύρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού του σχετικού με τη μεταφορά ζώων 2005, κανονισμός του 2005 και γίνεται αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας του κανονισμού. Επικριτική είναι η προσέγγιση του εισηγητού σα στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω τα πιο σημαντικά θέματα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, καταδεικνύει μία σειρά ε, δρομολογίων κατά τη μεταφορά των ζώων μεγάλης αποστάσεως, μεγαλύτερης από ό,τι αρχικά έχει προβλεφθεί, δηλαδή κατά την έκρηση του προπολογισμού, του κανονισμού. Γιατί τότε ε, είχε θεωρηθεί ότι θα περιοριστεί σταδιακά η απόσταση, η διενόμενη απόσταση. Αυτό ισχύει μόνο για τα άλογα. Ε, και για τα βοηθή οι αποστάσεις έχουν αυξηθεί κατά 7% ενώ για, τα, ε, για τους χείρους μέχρι και 70% έχουν αυξηθεί οι αποστάσεις, οι αποστάσεις, πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλο και περισσότερες είναι οι αποστάσεις τις οποίες, τις οποίες τα ζώα. Ενώ ο αρχικός στόχος του κανονισμού ήταν ξεκάθαρα να περιορίσει τα χιλιόμετρα που διανύουν τα ζώα. Πρώτον. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να μην έχει υπολογίσει πλήρως το κόστος των μεταφορών αυτών. Δηλαδή έχει λάβει υπόψη μόνο το κόστος για τον μεταφορέα. Ενώ θα έπρεπε να δούμε το κόστος συνολικά, περιβάλλον, ε, επιπτώσεις στους ε, πληθυσμούς που μένουν κοντά στους ε, δρόμους από τους οποίους παίρνουν τα, λεωφορεία, τα φορτηγά αυτά. Συνολικό κόστος λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην τιμή. Διότι δεν είναι ούτε στο συμφέρον του καταναλωτού, ούτε προς το συμφέρον του εκτροφέα του κτηνοτρόφου να ε, περνάει από αυτή την ε, μεγάλη διαδικασία από αυτές τις μακρές αποστάσεις που διανύει το ζώο. Είναι το πιο καλό προφανώς για όλους η σφαγή να γίνεται στον πιο κοντινό στον τόπο εκτροφής ε, χώρο και σφαγείο. Είναι προτιμότερο να γίνεται πρώτα η σφαγή και μετά να μεταφέρονται τα τεμάχια του κρέατος αντί να μεταφέρεται ζών, ζών το ζών και να ε, ταλαιπωρείται κατά την ε, διαδρομή αυτή. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία έχω υπογραμμίσει στην έκθεσή μου. Επίσης, ε, προσπαθούμε να ε, επισημάνουμε μία πρόταση μια αναθεώρηση του χρόνου ε, μεταφοράς στα ζώα που πηγαίνουν για σφαγή. διότι βλέπουμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τα ζώα εκτροφής, με τα ζώα μάλλον αναπαραγωγής ή ε, αγώνων ε, στα οποία ο ιδιοκτήτη, ή όποιος αναλαμβάνει να οργανώσει τη μεταφορά του έχει κάθε συμφέρον να τα προστατέψει για να έχουν καλές επιδόσεις στη συνέχεια. Ενώ τα ζώα που μεταφέρονται για σφαγή θεωρούνται μόνο αντικείμενα ε, για τον, από τον ε, ε, εκτροφέα, ιδιοκτήτη και ω εκ τούτου δεν υπάρχει επαρκής μέρημνα για την ευημερία του και τη συνθήκη μεταφορά. Επίσης, μπορέσαμε πρόσφατα να συλλέξουμε ε, υπογραφές με το ψήφισμα υπαριθμό 49 για τον περιορισμό του χρόνου μεταφοράς στις 8 ώρες. Και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να κατατεθεί μια πολύ πιο σαφή τροπολογία στο σχετικό κομμάτι. Θα πρέπει να μιλούμε για ένα σαφές όριο χρονικό, με βάση και τα όσα προτείνει το ψήφισμα υπαριθμών 49 διότι το Κοινοβούλιο έχει μέσω του ψηφίσματος αυτού ταχθεί ρητά υπέρ του περιορισμού στις 8 ώρες του χρόνου μεταφοράς των ζώων των ζώων. Και αυτό πρέπει να το αντικατοπτρίσει και η ε, έκθεση φαντάζομαι. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις βεβαίως. Εξαιρέσεις οι οποίες μπορεί να αφορούν ε, κάποιες περιοχές οι οποίες για λόγους γεωγραφικούς, για λόγους τοποθεσίας ε, είναι απαραίτητο να είμαστε πιο ελαστικοί, όπως για παραδείγμα οι νησιωτικές περιοχές, οι περιοχές οι οποίες είναι πολύ απομακρυσμένες. Αυτό ναι, αλλά με πάντα γνώμονα την ευημερία του ζώου. Δεν μπορεί το ζώο να το βλέπουμε σαν μία πηγή μόνο πρώτη ύλη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ζώα είναι όντα με αισθήματα και πρέπει να τα σεβαστούμε. Αυτά είναι λίγο πολύ οι ιδέες, αυτές ήταν οι ιδέες που μου οδήγησαν στη σύνταξη εκθεσίας μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Σα ενημερώνω όμω ότι η γραμματεία, όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων, έχει, έχει ε, καταρτήσει ένα πίνακα που θα σα δυναμηθεί μόλι τελείωσε και που καταγράφει τις ώρες ανά ζώου ή μάλλον τον αριθμό ζώων που μετακινούνται στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με το είδο, για να γνωρίζουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και πιστεύω να συμφωνεί και ο εισηγητής μαζί μου. 30 εκατομμύρια παραδείγματι είναι η οι χείροι ε, που ε, μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα πολλά εκατομμύρια τα βοηθεί και ούτω καθεξής. Παρακαλώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Βεβαίως και είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Μας το επενθύμισε και ο πρόεδρός μας μόλις τώρα. Πόσα πολλά ζώα δηλαδή μεταφέρονται οδικός στις χώρες μας. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα άκουσα. Όμως η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου συνηθίζει να επικρίνει την υπερβολική γραφειοκρατία και απαιτεί απλοποίηση και απαιτεί επίσης συχνά περισσότερη επικουρικότητα. Στην έκθεση όμως που έχουμε εδώ, κυρίως την παράγραφο 3 και την παράγραφο 10, εγώ καταλαβαίνω ότι αντίθετα ε, ζητούμε περισσότερη γραφειοκρατία και δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή πάνω σε αυτό. Οδηγία ή κανονισμό, ναι, μετά τα κράτη-μέλη πρέπει να το θέσουν σε εφαρμογή. Τον ελέγχει η Επιτροπή πώς θέτουν σε εφαρμογή τις αποφάσεις αυτές, τις πολιτικές αυτές, ε, οι χώρες είναι μια συνηθισμένη πολιτική. Δεν νομίζω ότι εμείς πρέπει ως προσανατολισμό να έχουμε την δημιουργία περισσότερης γραφειοκρατίας και περισσότερων εγγράφων. Τα μέσα πρέπει να τα έχουμε με τις υπάρχουσες δομές και να ελέγχουμε την εφαρμογή των νόμων. Επίσης, ο εισηγητής λέει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βρίσκει πληροφορίες από τα σφαγεία, από τις ε, ε, εταιρείες μεταφορών κτλ. με ερετηματολόγιο. Ναι, μα τις πληροφορίες αυτές Ακριβώς τις έχουν οι εταιρείε αυτές τα σφαγεία και τα λοιπά και είναι οι εθνικές διοικήσει οι οποίες πρέπει να πάνε και να επαληθεύσουν κατά πόσο είναι σωστές οι πληροφορίες που δίνουν ή όχι. Αλλά δεν μπορεί συστηματικά να πηγαίνουμε και να ρωτάμε εμείς όλους τους φορείς ενός κλάδου. Ευχαριστούμε Μισελ. Πρώτα κυρία Ρωμέ και μετά η κυρία Πέρες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση. Ένα γενικότερο πρόβλημα επισημαίνουμε ότι είναι ανεπαρκής, είναι μερική ατελής η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η εφαρμογή των υφισταμένων ε, νόμων. Αυτό είναι το πρόβλημα γενικότερα και δεν νομίζω ότι, χρεια... ότι είναι σκόπιμο να ε, τροποποιούμε νομοθεσία όσο δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμη την ουσιαστική υλοποίησή τη. Εδώ βλέπουμε να προτείνονται αλλαγέ ενώ δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμό. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Και καλό θα ήταν η ζήτηση να μην περιοριστεί μόνο στο χρόνο της μεταφοράς, γιατί καθίσατε πολύ επιφανειακή έτσι. Πρέπει να δούμε την ε, μεταφορά στο σύνολό της και τη γενικότερη ποιότητα της μεταφοράς, γιατί ε, προφανώς και έχει επιστημονικά ε, αποδειχθεί ότι είναι πολύ πιο ευχάριστο για τα ζώα να μεταφερόνται σε υψηλής ποιότητας, με υψηλής ποιότητας μεταφορικά μέσα και τρόπο μεταφορά. Επίσης θα πρέπει να αναλογιστούμε τι συνεπάγεται μια απόφαση που θα λάβουμε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίε απαραίτητα δεν, ε, δεν διαχειρίζονται απαραίτητα μεταφορικά μέσα ε, δικά τους και ως εκ τούτου πρέπει να εξαρτηθούν από την φόρτωση-εκφόρτωση σε περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα. Ο δε χρόνος μεταφοράς υπολογίζεται από την είσοδο στο μεταφορικό μέσο, από τη φόρτωση του πρώτου ζώου. Άρα ε, μπορεί Εάν κανείς έχει πολλά ε, ζώα και ε, βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή, να έχει εξαντλήσει το χρόνο της μεταφοράς, μόνο και μόνο φορτοεκφορτώνοντας τα ζώα του σε διαφορετικά μεταφορικά μέσα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ε, περιφέρειες στην Υπεθρό οι οποίες είναι κάπως πιο αποκομμένες από τα γενικά μέσα μεταφορές, από την άμεση δηλαδή φόρτωση ε, και παράδοση σε προορισμό. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και βέβαια πάντοτε με βάση επιστημονικά στοιχεία. Σημαντικό επίση είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον ε, κτηνοτρόφο να συμμετέχει ε, σε, μια, σε ένα ευρύτερο φάσμα επιλογής. Εάν τον περιορίσουμε μόνο σε ένα σφαγείο, γιατί θα του έχουμε περικόψει τόσο το χρόνο της μεταφοράς των ζώων, που δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να υπαχθεί σε ένα σφαγείο, δεν θα μπορεί να διαλέξει κάποιο άλλο, τότε ουσιαστικά του επιβάλλουμε ένα μονοπόλιο ως προς την προσφορά του προϊόντος του μόχθου του. Και αυτό ε, θα πρέπει φυσικά να μας απασχολήσει. Επίσης, όντως μπορεί ε, να προκαλεί άγχος, στρες η μεταφορά, αλλά δεν ε, είναι ο μόνος παράγοντας ε, άγχους. Δεν μπορεί δηλαδή ε, η διαδικασία της μεταφοράς και μόνο να υπολογιστεί ως παράγον ε, ε, άγχους, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συνθήκες, την ποιότητα δηλαδή των μεταφορικών μέσων, αλλά βέβαια και στη συνέχεια τις συνθήκες της ε, σφαγής, γιατί είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα με τις περιοχές και δεν μπορούμε κατά αποκοπή να δίνουμε λύσεις. Εάν πούμε λοιπόν ότι εισάγουμε το όριο των 8 ώρων και μετά ορίσουμε ότι μόλις περάσουν οι 8 ώρες πρέπει τα ζώα να, να εκφορτωθούν από το φορτηγό, να φεθούν σε έναν χώρο άγνωστο για αυτά, σε ένα περιβάλλον που δεν τους είναι οικείο. Αυτό επίσης σημαίνει σημαντικό στρες και άγχος για τα ζώα και πρέπει να το λάβουμε επίσης υπόψη. Γιατί ε, τότε βέβαια και αυτά ε, θα αισθανθούν άγχος, στρες, ε, δεν θα γνωρίζουν ε, τον χώρο, δεν θα μπορούν ενδεχομένως να τραφούν και να ποτιστούν σωστά. Και άρα το να επιβάλλουμε ε, κατά αποκοπή μια διάρκεια μεταφοράς 8 ώρες είναι σφαλμένη επιλογή, πιστεύω. Επίσης θα ζητούσα από τους αδέλφου οι οποίοι επιμένουν ανεφετέρου ε, στις 8 ώρες μεταφοράς τους καλώ να έρθουν να δουν τις διάφορες περιφέρειες για να δουν πώς μπορεί να κατασταθεί σφαγείο μέσα σε μια ακτίνα 8 ώρων μεταφοράς γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα βρεθούν οι συνθήκες για την κατασκευή ε, σφαγείου μέσα στο στην ακτίνα αυτή των οκτώ ωρών που να εξυπηρετεί τις μικρές ε, επιχειρήσεις, τις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις. Και αυτό βέβαια πάντα σε όρους διαφάνειας, όπως άλλωστε πατούμε και για την ε, μεταφορά των ζώων. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μπρίτα. Η μετά η Αντιπρόεδρος Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή που μας παρουσίασε τις κύριες ιδέες που περιλαμβάνει στην γνωμοδότησή του. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με την κυρία Ρέιμερς σε αυτά που είπε στην αρχή. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι η τρέχουσα νομοθεσία να διαθέτει όλα τα μέσα που χρειάζεται για να τίθεται σε εφαρμογή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε νέες προδιαγραφές, νέα νομοθεσία. Πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε να εφαρμόζονται τα όσα ήδη ισχύουν και συχνά δεν εφαρμόζονται. Εξού και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εφαρμόζονται τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τώρα, τα άλλα τα έχω πει και σε άλλες συζητήσεις. Εδώ θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Πρώτον, για το 8ωρο. Έλεγε ο συγητής ότι υπάρχει μια γραπτή δήλωση και ότι έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που πρέπει. Όντως, έτσι είναι. Και μια τέτοια πρωτοβουλία δεν λέω ότι δεν έχει σημασία, αλλά πρέπει και να προβληματιστούμε. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έχει νόημα η συζήτηση που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας τότε πρέπει να αλλάξουμε τρόπο εργασίας. Εγώ νομίζω ότι οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται μέσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να ακούγονται όλες οι απόψεις και μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Γιατί αλλιώς πολλές φορές θα έφτανε να μαζεύουμε υπογραφές για το ένα και το άλλο θέμα και να μην ερχόμαστε εδώ ποτέ να το συζητάμε και να προβληματιζόμαστε μαζί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω αυτό που έχω πει και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω και τώρα για το 8ωρο. Δεν υπάρχει νομική βάση που να λέει ότι αυτή είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση. Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα είναι θετικό για ορισμένα ζώα, σε άλλες περιπτώσεις θα είναι αρνητικό ή τέλο πάντων γιατί 8 και όχι 3 για το ένα ζώο ή για το άλλο. Δεν υπάρχει νομική βάση για αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να μου το εξηγήσει κάποιο ειλικρινά. Γιατί μιλάμε για 8 ώρες για τα ζώα που πηγαίνουν για σφαγή. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν λέμε ότι 8 ώρες πρέπει να είναι το ανώτατο για τη μεταφορά των ζώων, αυτό πρέπει να ισχύει για κάθε σκοπό, όχι μόνο για τη σφαγή. Γιατί τα τελευταία λεφτά της ζωής τους δηλαδή θέλουμε να τους κάνουμε χάρη και να τα μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο άνετα. Ας μου το εξηγήσει κάποιος, γιατί λέμε 8 ώρες μόνο για τα ζώα που πάνε για σφαγή. Και γιατί δεν υπάρχει νομική βάση. Αν ε, υπάρχει τότε θα έπρεπε να είναι για όλα τα ζώα ζώα και όχι μόνο για εκείνα που πηγαίνουν προς σφαγή. Έρχομαι και σε κάτι άλλο. Πολλές φορές αναφερθήκαμε εδώ στο κοινωνικό κόστος. Εγώ το καταλαβαίνω. Το οικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος, αλλά θα ήθελα κάποιο να μου εξηγήσει τι εννοούμε όταν μιλάμε για κοινωνικό κόστος. Αυτά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η συγκεκριμένη κατάσταση σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Τα περιφερειακά κράτη-μέλη επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τέτοιες πρωτοβουλίες για θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές. Τέλος, ελπίζω να μπορέσουμε στο χρόνο που μας μένει να υποβάλουμε ε, καλές τροπολογίες και έτσι να καταλήξουμε σε μία θέση ε, μέσω της οποίας θα βελτιώσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία για την μεταφορά των ζώων και για την καλή μεταχείριση των ζώων, έτσι ώστε όλοι να νιώθουμε ότι μας ικανοποιεί. Ευχαριστώ για την πρόεδρος Πόλσεν. Τώρα έχει το λόγο και μετά Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή, τον κύριο Βιτικόφσκι, για την τόσο καλή δουλειά που έχει κάνει. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και εκείνο το χειρίστηκε πραγματικά με ευαισθησία. Θίγει διάφορα θέματα, τα οποία ίσως δεν έχουμε συζητήσει πολύ. Το θέμα της υγείας, για παράδειγμα, ή το θέμα των ασθενειών που μπορεί να ξεσπάσουν κατά την μακρά μεταφορά ζώων, μακράς διάρκειας. Και υπάρχει κάτι εδώ με το οποίο νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Καλύτερα να μεταφέρουμε το κρέας για πολλές ε, ώρες παρά να μεταφέρουμε τέτοια τα ζώα τόσες πολλές ώρες. Και έπειτα πρέπει να δούμε αυτό το πολυδιάστατο θέμα που έχει να κάνει με τα σφαγεία. Ίσως εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια πρωτοβουλία από τη δικιά μας την ε, Επιτροπή. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι τις διαφορετικές διαστάσεις όσον αφορά τα σφαγεία στις χώρες μέλη, αλλά υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα εφόσον υπάρχουν δίκτυα μικρών σφαγείων. Και δεν είναι μόνο το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων, είναι και το θέμα και της ανάπτυξης, της υπαίθρου και της απασχόλησης. Άρα λοιπόν πρέπει να τη σκεφτούμε αυτή την δυνατότητα. Νομίζω ότι χρειάζονται καλύτερη έλεγχη και καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ίσως περισσότερους πόρους προκειμένου να μπορούν οι ίδιες οι χώρες μέλη να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση, να φτιάξουν κάτι σαν ένα FBI για παράδειγμα που να ελέγχει ε, την ε, κατάσταση. Στις χώρες μέλη δηλαδή να δημιουργηθεί μια τέτοια αρχή. Δεν ξέρω βέβαια από την άλλη οι ίδιες οι χώρες είναι υπεύθυνε για την δημιουργία τέτοιων αρχών και πολλές χώρες τις έχουν ήδη. Οπότε εμείς να εμπλεχτούμε, να αναμειχτούμε και να πούμε στις χώρες μέλη τι να κάνουν, δεν ξέρω. Πάντως αυτό το οποίο σίγουρα λείπει είναι μια δορυφορική, ένας δορυφορικός έλεγχος, κάποιο είδους GPS. Και έχουμε και ένα πολιτικό ζήτημα. Το οποίο όμως πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Γιατί έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές όσον αφορά την εκστρατεία για την μεταφορά των ζώων. Και γι' αυτό πρέπει μαζί να καταλήξουμε σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό με ισορροπία, να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή και την πραγματικότητα επιτόπου και ε, το θέμα της ε, μεταφοράς των οκτώρων Και εγώ υπέγραψα. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι η πιο ρεαλιστική εναλλακτική λύση, αλλά γι' αυτό προτείνω να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε ένα συμβιβασμό που να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα επιτόπου με τις γνώσεις που έχουμε και που έχει και ο συγγετής. Φαίνεται ότι οι 8 ώρες δεν είναι ότι το καλύτερο, γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη ζώων, διαφορετική ηλικία ζώων και επιπλέον πρόκειται για τις συνθήκες μεταφοράς ποιες θα είναι οι συνθήκες. Αυτές είναι αποφασιστική σημασία και όχι τόσο οι ώρες κατά τις οποίες μεταφέρεται το ζώο. Συνεπώς, οι καλές συνθήκες έχουν σημασία. Να έχουν νερό, καλό εξαορισμό, θέρμαση. Όλα αυτά είναι που πρέπει να σκεφτούμε και όχι μόνο να επικεντρωνόμαστε στον κανόνα του οχτάωρου. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί αυτή την πραγματικότητα εμείς καλούμεθα να διαχειριστούμε εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όμως, αυτό που άκουσα, κυρία Πόλσον, αυτό που άκουσα με οδηγεί να ζητήσω από τη Γραμματεία να μας δώσει πιο συγκεκριμένες ε, ενδείξεις, υποδείξεις, γιατί μεγάλο τμήμα, τουλάχιστον όσον αφορά το βοηδί, δεν είναι ζώα που μεταφέρονται για να σφαγιαστούν μετά. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών αφορά ζώα τα οποία ε, περνούν στην εκπάχυνση πρώτα. Για να σας δώσω το παράδειγμα της χώρας μου. 1,5 εκατομμύριο κεφάλια εισάγει η χώρα μου από τη Γαλλία και άλλα τόσα από τη Γερμανία. Νέα μοσχάρια τα οποία έρχονται, μένουν στην Ιταλία, τα παχαίνουμε εμείς εκεί και μετά πάνε στα σφαγεία. Άρα λοιπόν πάνε πολύ μακριά και σφαγιάζονται πολύ μακριά. Και τώρα το να σφάζει κανείς τα ζώα πολύ μακριά δεν είναι μόνο θέμα της μεταφοράς, είναι θέμα και οικονομικό. Δεν συμφέρει. Είναι σημαντικό λοιπόν η απόφαση που θα λάβουμε για την έκθεση Βοζιντουχόφσκι να βασιστεί στα νούμερα, στα στοιχεία που θα έχουμε, γιατί αλλάζουν πολύ τα πράγματα και η οπτική του προβλήματος αν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σμιτ. Και μετά Μάρτιν Όσνου. Uh, Σας ευχαριστώ. Εγώ θα εκφράσω ενδιαφέρον ως ε, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας στα ζώα. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για μια πολύ ισορροπημένη έκθεση, πράγμα που δεν ήταν εύκολο, είμαι βέβαιος, λόγω των πιέσεων που ασκούνται από όλες τις πλευρές. Και εμείς είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις στην ομάδα μου για αυτό το θέμα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία επί των οποίων συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι είναι ευκολότερο να μεταφέρει κανείς το κρέας αντί για τα ζώα και είναι και φθηνότερο. Τώρα το θέμα είναι μεταφορά προς το σφαγείο, είναι αυτό που είπε η κυρία Γκαρσία Περές. Γιατί μιλάμε για 8 ώρο όριο για τη μεταφορά προς το σφαγείο. Υπάρχει αίσθηση στο ευρύ κοινό πως τα ζώα που μεταφέρονται για σφαγή ε, τη διαφορετικές μεταχείρισεις από αυτά που πάνε για αλλού. Αυτή είναι μια αίσθηση, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει όντως, αλλά νομίζω πως αυτό οφείλονται αυτά όλα. Υπάρχει επιθυμία από τους λαούς μας να υπάρξει, να επιβληθεί κάποιο όριο. Θα πρέπει να δούμε αν είναι αυτό εφικτό και όντως επιθυμητό και πρακτικά και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις για μένα λοιπόν αυτή η έκθεση έχει βρει μια ανισορροπία ανάμεσα στο πρόβλημα το βασικό που είναι η καλύτερη εφαρμογή και την έλλειψη στοιχείων όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις κυρίως ε, στις τιμές των τροφίμων για τις προτάσεις αυτές που προχωρούν. Και σημειώνω την πρόταση αυτή που θα λέει ότι θα οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία. Το θέμα είναι ότι εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να εφαρμοστεί και σωστά. πρέπει να παρέμβουμε ώστε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν ε, μαρτυρίες, υπάρχουν μάλλον στοιχεία που δείχνουν ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο σε πολλά κράτη-μέλη. Τώρα, παράγραφος 5 λέει ότι χρειάζεται περισσότερα στοιχεία από την Κομισιόν, όχι μόνο για την καταμέτρηση και πού πάνε και πού έρχονται, από πού έρχονται τα ζώα, αλλά κυρίως για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των δυνητικών αποφάσεων που λαμβάνουμε εμείς εδώ για το κόστος του κρέατος και συμφωνώ και με την κυρία Ράιμερς που είπε ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς ως ένωση εν γέννη, ότι δηλαδή όσα περνάνε από εδώ θα πρέπει να είναι συνεπείς με το άλλο νομοθετικό σώμα. Και έχει δίκιο η κυρία Πόλσον ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου και το να δίκτυο μικρών σφαγείων θα ήταν κάτι το επιθυμητό, όμως υπάρχουν προβλήματα με άλλα κομμάτια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αυτό το καθιστούν δύσκολο στην εφαρμογή. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα στη Σκωτία που είχαμε διάφορα μικρά σφαγεία που έπρεπε να κλείσουν λόγω των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και γιατί δεν έβγαιναν οικονομικά. Υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις λοιπόν ε, πορεών από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει εμείς ως νομοθέτες να ε, προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά που έχουν εντοπιστεί. Τώρα για την παράγραφο 19. Πολύ αμφισβητήσιμο ε, αυτή η διατύπωση. Αυτό που ζητά είναι να εξετάσουμε παρεδέρω την ανάγκη σε αυτού του ορίου. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για το κατά πόσο είναι εφικτό αυτό ή όχι. Μπορούμε να δούμε όμως το κατά πόσο επιθυμούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια προσέγγιση unisex για όλους η ερώτηση του κατά πόσο το οκτάωρο είναι κατάλληλο για κάποια είδη σε σχέση με κάποια άλλα, τις συνθήκες για τα κάποια ζώα. Σε κάποια μέρη της χώρας μας, κάτι τέτοιο δεν γίνεται και θα σήμαινε την κατάργηση της εκτινοτροφίας σε μεγάλα κομμάτια της χώρας μου. Φαντάζομαι το ίδιο και για άλλες χώρες. Και αυτό δεν είναι καλό ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την ανάπτυξη, ούτε και για τους λαούς μας εν γέννη. Νομίζω λοιπόν πως τελικά βρήκε μια υγιή ισορροπία ο εισηγητής, θα κάνουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι θέλουμε να γίνει και να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις επιπτώσεις των αποφάσεών μας δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων εδώ σε αυτό το θέμα και χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Μάρτιν Όσλινγκ και μετά η κυρία Γέγκλε. Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Πιστεύω ότι αυτό το 1 εκατομμύριο ε, υπογραφές ε, της ε, εκστρατείας συλλογής νομίζω πρέπει να τις υπολογίσουμε με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα και δεν μπορούμε να ξεκινάμε μια συζήτηση λέγοντας προκαταβολικά τι δεν δεχόμαστε, τι δεν πάει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να αποφεύγουμε στις μεταφορές των ζώων. Το να αυξηθούν μέσα σε τέσσερα χρόνια κατά 70% οι μεταφορές χείρων στην Ευρώπη προφανώς είναι λάθος, προφανώς δείχνει ότι κάπου έχουμε κάνει λάθος. Ας μην ε, γελιοποιούμαστε. Η κατάσταση στη Γερμανία βεβαίως μπορεί να είναι διαφορετική ως προς τα σφαγεία, γιατί υπάρχουν τα μεγάλα σφαγεία, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και ανάλογα και ο εκτροφέας αντιμετωπίζει τη σχετική δυσκολία στην πρόσβαση στο σφαγείο. Από την άλλη θα πρέπει να προωθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο περιφερειακές τομές και με τους δύο πυλώνες ε, που έχουμε στη μας θα μπορούσαμε ενδεχομένω να προωθήσουμε αυτή την ιδέα της περιφερειακής, του περιφερειακού δικτύου σφαγείων ώστε να μην ε, συνεχιστεί αυτός ο φαύλος κύκλος, να διαρρήξουμε το φαύλο κύκλο. Δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος ένας κτηνοτρόφος ε, να ε, μεταφέρει τα ζώα του από τη Σουηδία μέχρι το Σλέσφικ Χολστάιν για να τα σφάξει. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και βέβαια στην αναπαραγωγή, στην εκτροφή αλλά και στη σφαγή πρέπει να έχουμε στο δυνατόν πιο μεγάλη, ε, πιο μεγάλη προσοχή στην ευημερία του ζώου και οικονομία στον χρόνο μεταφοράς. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να ε, βάζουμε στον ίδιο κουρβανά τα ζώα εκτροφής με αυτά που ε, μεταφέρονται για λόγους αγώνων, παραδείγματι αναπαραγωγής. Φανταστείτε ένα άλογο για το οποίο θα απαγορευτεί η μεταφορά πάνω από 8 ώρες διάρκειας και δεν θα μπορεί να ε, πάει να συμμετάσχει σε αγώνες σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης. Από την άλλη έχουμε δει τις εικόνες, τις δυσάρεστες συνθήκες μεταφοράς ζώων προς σφαγή. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση. Και επίσης Νομίζω ότι ό,τι ωραίες διατάξεις και να εισάγουμε, ό,τι ωραίες και καλές προθέσεις να έχουμε, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι στην εφαρμογή της νομοθεσίας, αν δεν υπαλληθεύεται ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας, τότε δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν, η κυρία Γέγκερ και μετά ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. με παραξενεύει το γεγονό ότι είμαι υποχρεωμένη να ομολογήσω πως συμφωνώ σε πολλά σημεία με τον κύριο Χόισλινγκ και το ομολογώ εγώ ίδια πρώτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι μια ισορροπημένη έκθεση. Αλλά όπως είπε, δεν ενδιαφέρει το Γεωργό πόσα... Αλλά είπε ότι δεν ενδιαφέρει το Γεωργό ε, ζώα μεταφέρει. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό, εάν το κατάλαβα σωστά δεν του είναι αδιάφορο του οδηγού, του ε, γεωργού, του κτηνοτρόφου πόσα ζώα θα μεταφέρει. Αλλά έχει ε, προκύψει ως συνέπεια των διαφορετικών νομοθεσιών που ισχύουν στα κράτη-μέλη ότι πολύ συχνά τα κρατά ε, ζώα ανάλογα με την κατηγορία ή τη χρησιμότητα που έχουν για τον εκτροφέα τους αν πρόκειται για ζώα για αγώνα, αν πρόκειται για ζώα αναπαραγωγής, αν πρόκειται για ζώα που πάνε στη διασφαγή αναλόγως και με φθήνουσα βέβαια σειρά ε, έχουν και ε, τις συνθήκες μεταφοράς. Δηλαδή τα ζώα πάνε για σφαγή έχουν δυστυχώς τις χειρότερες συνθήκες μεταφοράς. Για το χρόνο μεταφοράς μπορούμε να συζητήσουμε και το οκτάωρα και τις συνθήκες ή τις ώρες μεταφοράς, ε, φόρτος εκφόρτωσης, αναλόγως με την περιοχή αν χρειάζεται να παρατείνουμε τη διάρκεια της μεταφοράς λόγω κάποιων διαζουσών συνθήκων. Επίσης για τα σφαγεία και τα περιφερειακά δίκτυα σφαγείων. Έχω άλλωστε επισημάνει τις θέσεις μου πιστεύω και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Πρέπει νομίζω και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και άλλες επιτροπές, να το δούμε το θέμα πιο γενικά, διότι δεν πρέπει να έχουμε υπόψη, ε, δεν πρέπει να κατηγορούμε μόνο τον ε, ε, εκτροφέα ο οποίος δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές ή όλους αυτούς που ε, εργάζονται γύρω από ένα σφαγείο. Τα μικρά σφαγεία, τα μικρά περιφερειακά σφαγεία, η δική μας νομοθεσία τα έχει οδηγήσει σε κλείσιμο και άρα χρειαζόμαστε διαφορετικές δομές, περιφερειακές δομές, ε, συνθήκες μεταφοράς κατάλληλες για τα ζώα αυτά για εκτροφή και βέβαια υπολογιζομένου και του κόστου της μεταφοράς όταν έχουμε να κάνουμε με τη μεταφορά εκατομμυρίων ζώων. Βεβαίω οι μεταφορές μπορεί να λέει θα προτιμούσα αυτό, εκείνο ή το άλλο να είναι καλύτερα ε, σχεδιασμένα, αλλά ε, δεν μπορεί παρά να εφαρμόσει την νομοθεσία την οποία εμεί έχουμε εισαγάγει και αυτό ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε. Και επίσης έλεγχος και εφαρμογή τη νομοθεσία. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα και όχι το να εισαγάγουμε περισσότερε διαδικασίες και γραφειοκρατία. Έτσι πρέπει να προβληματιστούμε και σε αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε, γιατί το πρόβλημα υπάρχει στην Γερμανία, φαντάζομαι, όχι μόνο. Είναι οι δομές των μεταφορών και οι συνθήκες μεταφοράς των ζώων και έτσι ενώ τα ζώα τα ίδια, τα βοηδή φερρυπέν έχουν μεγαλώσει, είναι πιο μεγάλα για λόγους ε, εκτροφής, ευγονικής και το οι συνθήκες που έχουν προβλεφθεί αφορούν άλλα μεγέθη ζώων, άλλες διαστάσεις ζώων και δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί, ενώ θα έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Και γι' αυτό θα ήθελα και να έχω μια πιο επακριβή συζήτηση για τα νούμερα. Μήπως θα ήταν πρόεδρε να έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε μια γενικότερη συζήτηση, όχι μόνο τις 8 ώρες, τον τρόπο μεταφοράς κλπ. Να μιλήσουμε εν γέννη για συνθήκες, μεταφοράς και άρα θα έπρεπε ή δυνατόν, ή δυνατόν να αναβάλουμε για λίγο την έκθεση, να τη δώσουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και με πολύ πιο επακριβή στοιχεία ποια είναι η συνθή, κατάσταση που επικρατεί και πού θέλουμε να πάμε. Και βέβαια θα δώσουμε και το σχετικό περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει τι προτάσει τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελίζα. Πρέπει να επιλέξουμε την πιο αποτελεσματική στρατηγική. Τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ε, με το ότι ο εισηγητής ε, προβλέπει το θέμα της γεωγραφίας εδώ. Ο κ. Σμίτη τόνισε την ε, Σκοτία, έχουμε τα Highlands, έχουμε νησιά, Μεγάλε αποστάσεις. Πριν από 20 χρόνια επευλήθη δρακόντια νομοθεσία για τα σφαγεία και το αποτέλεσμα ήταν στον Ηνωμένο Βασίλειο καταλήξαμε στο να έχουμε πολύ λίγα και τεράστια σφαγεία. Αυτό σημαίνει πως αν ε, προχωρήσουμε σε αυτή τη γραμμή, ότι δηλαδή τα ζώα πρέπει να πάνε στο πιο κοντινό σφαγείο, θα δημιουργηθεί αμέσως ένα μονοπόλιο. Διότι αν μπορεί κανείς να πουλήσει μόνο σε ένα σφαγείο, εκείνο μπορεί να, να ορίσει τις τιμές και αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα πάνε ε, εκεί και θα φύγουν από τις αγροτικές περιοχές. Ελπίζω πως αυτό θα φύγει από εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα εξάλλου αν επιβαλόταν ο ισχύων νόμος. Και αν δούμε και άλλους νόμους για την ευημερία, για τις κλοβούς, ε, ε, δεν έχουμε πολύ καλό ρεκόρ όσον αφορά την επιβολή νομοθεσίας. Ε, νομίζω πως δεν έχει νόημα να φτιάχνουμε ακόμα πιο αυστηρούς νόμους όταν τους ισχύοντες δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε. Επίσης ανησυχώ κάπως για το πότε ξεκινά η ημέρα μεταφορών. Εγώ όταν φορτώναμε φορτηγά, ο οδηγός και εγώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά σε κάτω από μια ώρα. Μιλάμε για τεράστια φορτηγά. Πρέπει να πα σιγά σιγά. Κάποιε φορέ τα ζώα δεν έχουν καμιά όρεξη να μπουν μέσα στα φορτηγά. Ιδιαίτερα αν είναι με γεμάτα τα στομάχια. Λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να πάνε με γεμάτο στομάχι μέσα στο φορτηγό. Είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει γιατί ακριβώ αρχίζει αρχίζουν να μυρικάζουν τη στιγμή που μπαίνουν μέσα στο φορτηγά. Ε, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ, πολύ, πολύ χρονοβόρο το να μπουν μέσα στα φορτηγά και μετά πάλι δεν έχουμε μια όρεξη να βγουν από τα φορτηγά. Αυτό το πολύτιμα φορτία δε, δεν, ε, δεν θέλει κανείς να τα τα χειρίζεται για να χάνει λεφτά. Είναι πολύτιμα. Κανένας δεν θέλει να βγαίνουν νεκρά ε, βόδια από το φορτηγό στο σφαγείο. Είναι βάζει τον ε, μεταφορέα σε δύσκολη θέση και είναι και ζημιά. Βέβαια. Ευχαριστώ. Μάριν Μαγκίνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου, γιατί τρέχω ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και την δική μα εδώ τη Γεωργία. Είναι σημαντική η συζήτηση όμω Νομίζω ότι αυτό που είπε η κυρία Γέγκλε, να δώσουμε περισσότερο χρόνο να το σκεφτούμε, είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί αναφέρθηκαν θέματα από όλους για την ελέγχου. Με παραπάνω νομοθεσίε δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί και η κατάσταση για τα ζώα. Εάν βάλουμε αυτόν τον κανόνα των 8 ώρων, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τις 8 ώρες και όχι με τις 10 ώρες ας πούμε. Πρέπει όλα αυτά να τα ξαναδούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο στη συζήτηση αυτή. Επίσης η Ευρώπη έχει μετακινηθεί έχει, έχει μάλλον απομακρυνθεί από τα μικρά σφαγεία. Σε όλα τα κράτη-μέλη έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, μεγαλύτερες ε, ε αποστάσεις μέχρι τα σφαγεία και βέβαια θέματα μονοπωλίων. Πρέπει και αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Μεγαλύτερη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή είναι για τα άλογα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν είναι το υψηλότερο, ε, είναι μάλλον το ψηλότερο επίπεδο δεν μιλάμε για εκείνα τα άλογα πολυτελείας που είναι, ταξιδεύουν με όλα τα κομφόρ όπως και εμείς όταν ταξιδεύουμε, αλλά για το χαμηλότερο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα σκεφτούμε και παρακαλώ τον εισηγητή να σκεφτεί και να σημειώσει τα σχόλια των συναδέλφων και να τα συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Και τώρα ο κύριος Μάκενταϊρ. η κυρία συγγνώμη Μάκενταϊρ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Επειδή είμαι και εγώ μέλος της ECR, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βόση Χόφσκι για τη δουλειά που έκανε σε αυτό το ενέκθεση. Νομίζω πως κατάφερε να συγκεντρώσει τη συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε όλοι ευαισθησία όσον αφορά το θέμα της ευημερίας των ζώων. Την περασμένη φορά που το συζητήσαμε είχα πάρει το λόγο και απλά θα ήθελα να επαναλάβω πως και ξέρω πως αυτό επηρεάζει και άλλες χώρες, αλλά στη δική μου περιοχή τα μικρά σφαγεία έχουν κλείσει λόγω της νομοθεσίας της Ένωσης ότι δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς νομοθετούμε λόγω των συνεπειών που καμιά φορά δεν είναι ηθελημένες. Ε, ανησυχούμε πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο για την μεταφορά αλόγων κούρσας και νομίζω πως αυτό είναι το συγκεκριμένο ζώο που έχει δημιουργήσει τις μεγαλύτερες ανησυχίες και, τα και που κινεί τα μεγαλύτερα αισθήματα. Θα πρέπει ίσως ε, να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα ζώα και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρονται τα ζώα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μεταφέρονται αδύναμα ή τραυματισμένα ζώα. Και αυτό κάπως θα πρέπει να τονιστεί. Εν γέννη όμως υποστηρίζω το είναι έκθεση. Ωραία. Τώρα θα ζητήσω από, τον, από τους εκπροσώπους της Επιτροπής αν θέλω να πάρω το λόγο. Sì, prego. Allora, e poi... Γκαμπινέλη, μάλιστα. Ζεβόσκι. Prego, Commissione. Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τη συζήτηση και προφανώς τον κύριο Φωσιχόφσκι για την έκθεση που παρουσίασε. Η Κομισιόν με μεγάλο ενδιαφέρον δέχεται το αίτημα για μια συζήτηση με περισσότερα στοιχεία και με την εφαρμογή του κανονισμού που προβλέπει διάφορες διατάξεις για να βελτιώσει την ποιότητα των μεταφορών. Εν συντομία θα μπορούσα να πω ότι η θέση της Κομισιόν είναι και μάλιστα έχουμε παρουσιάσει και έκθεση για το θέμα αυτό που λέει ότι η υπόθεση του χρόνου μεταφοράς είναι μόνο μία παράμετρος όσον αφορά την ποιότητα και τις επιπτώσεις ε, στην ευημερία των μεταφερόμενων ζώων. Και η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων στην έκθεσή του της, συγγνώμη, τόνισε ότι πέρα από το θέμα της διάρκειας ε, το θέμα είναι η ποιότητα, δηλαδή οι θερμοκρασίες και η ε, ένταση της μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε συγκεκριμένες προτάσεις για να βελτιώσουμε τους ελέγχους και την ανιχνευσιμότητα στα κράτη-μέλη. Θα σας ενημερώσουμε και για την κατάσταση των εργασιών μας ε, που είναι υπό εξέλιξη και σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας και τη συνεργασία σας. τα ευχαριστώ την Επιτροπή και δίνω και πάλι το λόγο στον Αντιπρόεδρο Φωζηγόφσκι ε, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της συζήτησης που μόλις έγινε, τη σημασία των παρεμβάσεων που έγιναν και τις πρότασεις που έκανε η Ελίζα Μπεθ καθώς και της προσοχής που πρέπει να δώσουμε στις προθεσμίες για την έγκριση αυτής της έκθεσης. Σημασία δηλαδή το να έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις για συγκεκριμένα ζώα, γιατί τα άλογα αναμφίβολα είναι διαφορετικά και θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση αυτή καθώς και όπως είπαμε αριθμητικά στοιχεία για να αξιολογήσουμε ανάμεσα στις μεταφορές ζώων που πάνε για σφαγείο και μεταφορές ζώων που είναι σε εκπάχυνση, που για ορισμένα είδη όπως τα βοήδη είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ο κύριος Σιγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις πρόσθετες ε, πληροφορίες και τις θέσεις που εκφράστηκαν. Ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά. Βεβαίως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο προήμιο τα σχετικά με, το, με την έκταση του φαινομένου της με των μεταφορών, το γεγονός δηλαδή ότι έχουν αυξηθεί οι μεταφορές και η διάρκεια. Ε, δεν τα είχα υπόψη, με ευχαριστώ πολύ, θα τα λάβω υπόψη, θα τα συμπεριλάβω στο κείμενο. Και Κυρίες και κύριοι, πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε τα θέματα των μεταφορών ζώων για αγώνες τα οποία έστω και αν δεν τιμώνται με μετάλλια χρυσά, είναι επάξια, είναι Ολυμπιονίκες. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τα ζώα που μεταφέρονται για αγώνες ή για αναπαραγωγή, αλλά για αυτά που πηγαίνουν στα σφαγεία. Και δεν είπα, κυρία Γέγκλε, ότι δεν ενδιαφέρει τον κτηνοτρόφο ο τρόπο ε, της μεταφορά ε, που επιλέγεται. Μπορεί τώρα να μην είμαι εγώ ο ίδιος κτηρινοτρόφος, αλλά έχω εργαστεί παλαιότερα όταν ήμουν νεαρός, δούλευα στο ε, αγρόκτημα των γονέων μου. Άρα προφανώς και ξέρω ότι τον ενδιαφέρει τον Γεωργό. Ο μεταφορέας δεν ενδιαφέρεται για την εφημερία των ζώων. Διότι ε, όταν ένα ζώο μεταφέρεται γιατί θα, θα χρησιμοποιηθεί σε αναπαραγωγή πρέπει να φτάσει υγιές. Ενώ όταν ένα ζώο μεταφέρεται μόνο για να μπει στο σφαγείο, ακόμα και αν φτάσει με σπασμένο πόδι στο τέλος διαδρομής, δεν ε, έχει σημασία ότι ή άλλος κατάληξη του θα είναι η ίδια. Ε, και βεβαίως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές το 1 εκατομμύριο υπογραφές που συλλέχθηκαν κατά την εκστρατεία με το ψήφισμα Συμφωνώ με τους αδέρφους που λένε ότι δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την ε, ανησυχία του κοινού. Ε, είναι τραυματικές αυτές οι καταστάσεις, έστω και αν σημειώνονται κάποιες βελτιώσεις στο τομέα των μεταφοράς των ζώων, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις κακές πρακτικές. Επίσης, ε, κάποιοι μιλούν για προβλήματα σχετικά με τα σφαγεία. Εγώ, καθώς έχω ανεκτό μυαλό, αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο, στη μεταφορά, αλλά, όπως λέω άλλωστε και στην παράγραφο υπαριθμών 8 της εκθεσεώς μου, πιστεύω ότι θα πρέπει να επαληθευτεί εν γέννη η πολιτική η γεωργική και ε, να επιδιώξουμε να στηρίξουμε περιφερειακά, μικρά δηλαδή, ε, σφαγεία, ίσως μέσω του δεύτερου πυλώνα. Θα πρέπει να προσφερθεί φερρυπίν οικονομική στήριξη σε σφαγεία που φερρυπίν δεσμεύονται να ε, προμηθεύονται το κρέας από ή τα ζώα καλύτερα από ε, κτηνοτρόφους της περιοχής. Αυτό με μια τέτοιου τύπου δέσμευση μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα για βελτίωση της στον των ζώων. Αν και γνωρίζω από την Πολωνία τουλάχιστον ότι η εκμεταλλεύση είναι επιτοπλίστων μεγάλης έκτασης. Επίσης, δεν ξέρω σωστά, να μην κατάλαβα καλά την ε, παρέμβασή σας, αλλά θεωρώ ότι εκεί όπου διαπιστώνονται μονοπόλια, όσο ε, λιγότερα είναι τα σφαγεία, όσο μικρότερη δηλαδή είναι η επιλογή για τον κτηνοτρόφο, τόσο πιο δύσκολη είναι η θέση του, τόσο ενισχύεται το μονοπόλιο δηλαδή. Ενώ αν έχουμε περισσότερα σφαγεία στη διάθεση του κτηνοτρόφου, προφανώς μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός πιο ικανοποιητικά. Εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι, εγώ προσπάθησα στην έκθεσή μου να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν ε, πιο ε, πολλά, ε, όσο πιο πολλές ε, διαφορετικές πτυχές μιας ε, λύσης η οποία θα είναι η καλύτερη για τα ζώα. Ίσως οι 8 ώρες να είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση στο χώρο των μεταφορών. Πάντω δική μου πρόθεση δεν ήταν, κύριε Ντόντα, να ενισχυθεί η γραφειοκρατία. Δεν υποστηρίζω περισσότερη γραφειοκρατία. και εκεί όπου γίνεται λόγος για εξειδικευμένη υποστήριξη, εξειδικευμένα ελεκτικούς θεσμού στα κράτη-μέλη, στο σημείο 3 της εκθέσεως που ανέφερε και η κυρία Πόλσεν, θα ήθελα να πω ότι εμείς στην Πολωνία δεν έχουμε τέτοιους θεσμούς ελέγχου που θα εξασφάλιζαν επαρκώς την προστασία ή κατά κύριο λόγο την προστασία των ζώων. υπάρχουν οι υπηρεσίες εκτινοτροφικές οι οποίες μεριμνούν ε, για το θέμα αυτό, αλλά παρεμπιπτόντως. Και έτσι, εάν εισάγονται τόσες διατάξεις για την ευημερία των ζώων ή μη τι άλλο, θα έπρεπε να έχουμε κατάλληλα σώματα ελεγκτικά στα κράτη-μέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επαληθεύουν την ουσιαστική την σωστή εφαρμογή τήρηση των διατάξεων. Επιτρέψτε μου κλείνοντα να πω ότι στην κατάρτιση αυτή τη έκθεση ο δικό μου είχα και την προσωπική μου ευαισθησία αλλά και ε, μελήματα οικονομική τάξεω. γιατί φερειπίν ε, πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλο όγκο μεταφορών ε, από την Πολωνία στην Ιταλία και πολλοί μπορεί να διαμαρτύρονται και να λένε ότι οι Πολωνοί κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να πολλούνται τα ζώα του για ε, σφαγή στην Ιταλία και έτσι να μεταφέρουν τα ζώα αυτά από την Πολωνία μέχρι την Ιταλία. Ε, ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι οι προτάσεις που κάνω δεν υπαγορεύονται από την ε, πρόθεση να υποστηρίξω ή να ε, ωφελήσω περισσότερο τους Πολωνούς γεωργούς. Γιατί τόσο ο Πολωνός γεωργός όσο και ο Ιταλός καταναλωτής έχουν συμφέρον το κρέας το οποίο θα πουλήσουν ή θα καταναλώσουν να είναι να έχει παραχθεί στο δυνατόν πιο κοντά στον ε, χώρο διαβίωσης εκτροφής του ζώου. Επίσης δεν θέλω να επισημώνω ότι έχουμε υιοθετήσει την ε, ε, δήλωση παριθμών 49, την έχουν υπογράψει πολλοί βουλευτές και δεν μπορούμε να εκδίδουμε αντιφατικά με προηγούμενες δηλώσεις κείμενα. Ο κύριος ε, Βιζόφσκι, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους για τον ε, χρόνο που μου προσφέρατε για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλή εργασία σας εύχομαι, κύριε Αντιπρόεδρε Φωσιγόφσκι. Ευχαριστώ όλους. Ε, θα ξαναρχίσουμε τη συνεδρία μας στις 3. Σας θυμίζω ότι στις 3 ε, θα έχουμε μια σημαντική παρουσία του συναδέλφου Ράιμερ Κόγκη και Κάλφιν για το οικονομικό ζήτημα, γι' αυτό σας ζητώ να είστε παρόντες. Μάρια, ήθελες να παρέμβεις? Όχι. Ωραία. Εντάξει, γεια σας. Καλή όρεξη.